Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση και έχω να σας κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Αν δείτε λιγάκι την ε, ημερήσια διάταξη, μισό λεπτό λέει ο Πρόεδρος, Υπάρχουν κάποιες ε, αλλαγές και θα ήταν καλό ε, αν και εσείς λέγατε τη γνώμη σας επ' αυτών. Δηλαδή, τα σημεία 4 και το 11 αναβάλλονται για την επόμενη συνεδρίαση και υπήρξαν ε, κάποιες ε, τεχνικές δυσκολίες στην έκθεση της συναδέλφου Χάκιν. Άρα ούτε το 4 θα εξετάσουμε, ούτε το 11 στην ψηφοφορία. Άρα δηλαδή διαγράψτε τα, πάει το 4, πάει και το 11. Και Υπάρχει μία αλλαγή στην ημερήσια διάταξη, δηλαδή το 20 και το 21 θα ε, τα εξετάσουμε μετά το 12. Το 20 και το 21 θα πάνε αμέσω μετά το 12. Για το 13, αυτό θα το εξετάσουμε μετά το 15 και το 19 μετά το 16. Αυτά είχα να σας πω. Τώρα η δεύτερη παρατηρήσει που θέλω να κάνω. Εντάξει, όλα αυτά είναι τεχνική φύση θέματα, δεν είναι σημαντικά και επειδή είμαστε ευέλικτοι, νομίζω δεν ε, υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά την ε, Annual Interpretation, εκεί κανεί ε, δεν ζήτησε την γραπτή μετάφραση και γι' αυτό δεν έγινε. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι είναι προφανές ότι μας ακούνε εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών γιατί η συνεδρίαση μας μεταδίδεται μέσω Web TV. Κατόπιν τούτου, να ξέρετε, οι συνάδελφοι που πάντα έχετε πολύ ε, αποτελεσματικές ε, παρεμβάσεις, να γνωρίζετε ότι σας παρακολουθούν εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίων πολιτών. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης που είναι τα πρακτικά της 29ης και 30ης Μαΐου και 19 και 20 Ιουνίου. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει ε, καμία παρέμβαση, ε, νομίζω εγκρίνονται τα πρακτικά. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 4. Πάει αυτό, το είπαμε, άρα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για τις υπόλοιπες εκθέσεις. Ο συνάδελφος Κάζα έχει αρρωστήσει, αλλά ο Hans Becker, ε, που είναι πολύ δυναμικός, θα λάβει το λόγο. Χάντς, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας διαβάσω την σύντομη έκθεση του συναδέλφου Κάζα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σαφές πλαίσιο για να καθοδηγήσει τις πολιτικές ενέργειας και κλίματος μέχρι το 2020. Αυτό συμπεριλαμβάνει διάφορους στόχους πολιτικές και συμπεριλαμβάνει και η στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Τώρα ήρθε η στιγμή να σκεφτούμε για ένα νέο πλαίσιο 2030 για τις πολιτικές ενέργειας και κλίματος. Αυτή η γνωμοδότηση θα τροφοδοτήσει τη διαδικασία διαβούλευσης ομοδότηση βασίζεται σε αντιστοιχεία δεξιοτήτων, προετοιμασία του εργατικού δυναμικού και οικονομική στήριξη για αλλαγή στην ε, βιομηχανική διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Χάιντς, ε, και για τα θαυμάσια αγγλικά σου, που είναι μία από τις βασικές σου ικανότητες. Η συνάδελφος Κρεβέτη είναι σκιώδης εισηγήτρια για τους σοσιαλδημοκράτες. Μην... Έχετε το λόγο. Θα ήθελα ξεκινώντα θα να απευθύνω τις ευχές μου στον ε, συνάδελφο Κάζα και σαν σκιώδης εισηγήτρια εγώ ε, συνέταξα διάφορες τροπολογίες και αυτό τον οργιακό παράγοντα τον έλαβα πραγματικά υπόψη μου γιατί σημαίνει θέσεις εργασίες αλλά ταυτόχρονα και την ανάγκη να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Ειδικά θα ασχοληθώ με τις πηγές για τα green jobs και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί, γιατί εκεί αυτές θα πρέπει να προσέξουμε Επίσης ασχολήθηκα με το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και να τις εγγυηθούμε πραγματικά αυτές τις συνθήκες εργασίας και ακόμα καινούρια στοιχεία για αυτές τις πράσινες θέσεις εργασίας γιατί είναι ειδικέ εργασίες επαναλαμβάνω και υπάρχουν όλο ένα και περισσότερο δυνατότητες που ανοίγονται στα πλαίσια αυτά. Είναι σημαντικό γιατί γιατί νέος κόσμος που είναι ιδιαίτερα ενεργός, δραστήριος όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος ενδιαφέρονται για αυτές τις πράσινες θέσεις εργασίες. Α, λοιπόν, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. Είναι καλή αυτή η έκθεση λοιπόν και σας ευχαριστώ. Και είναι και σημαντική. Ευχαριστούμε πολύ από τους σκιώτες. Θέλει κανείς άλλος το λόγο. Από ό,τι βλέπω όχι ε, κάποιος άλλος που να θέλει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρο Μπαρόσο στην ομιλία του για την κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ότι η Κομισιόν του Επόμενου Μήνε θα παρουσιάσει πιο συγκεκριμένε προτάσει ε, για το πλαίσιο για το 2030. Επομένω, οι επόμενοι μήνε είναι κρίσιμοι για να καθορίσουμε ένα φιλόδοξο πλαίσιο βάσει των τριών πυλώνων ε, τη ενεργειακή και κλιματική πολιτική, ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια του εφοδιασμού και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ξέρετε ότι έχουμε υιοθετήσει ε, μια σχετική πράσινη βίβλο και επομένως είναι ουσιαστικό να έχουμε μια πρώμη συμφωνία για το πλαίσιο για να έχουμε μακροπρόθεσμη ασφάλεια και όραμα για τους επενδυτές τους και τους πολίτες. Ε, εδώ θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση του κύκλου του μακροπρόθεσμου για τις επενδύσεις και να έχουμε ασφάλεια για τις επενδύσεις. Επίσης, είναι ζωτικό το πλαίσιο για να καθορίσουμε μια νέα θέση εν ώψη διεθνών διαπραγματεύσεων στο Παρίσι το 2015. Και τέλος, το πλαίσιο 2030 είναι σημαντικό για να υποστηρίξει την ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα που προωθεί την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και δημιουργεί θέσεις εργασίας σε όλα τα κράτη-μέλη. Έτσι, η Κομισιόν θα ήθελα να καλωσορίσω τη συζήτηση στην Επιτροπή Απασχόλησης και την συνεισφορά αυτής της Επιτροπής σε όλη τη συζήτηση. Για να ολοκληρώσω, θέλω να δηλώσω ότι μέχρι τώρα ε, καλωσορίζουμε τη συνεισφορά του κοινωνικού πανέλ ε, στη συζήτηση και η κοινωνική διάσταση θα έχει μεγάλη βαρύτητα στον προβληματισμό της Κομισιόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλο το λόγο, άρα η διορία είναι 24 Οκτωβρίου στις 12 η ώρα και μετά προβλέπεται η ψηφοφορία το Δεκέμβρη και την ε, Ολομέλεια, ε, την πρώτη Ολομέλεια του 2014. Κατόπιν θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα δράσης ε, για την Χαλιβουργία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ευχαριστώ γιατί η Επιτροπή μας αποφασίζει έτσι να τοποθετηθεί σχετικά με τη χαλιβουργία και με τη γνωμοδότησή μας. Με τη γνωμοδότηση δε αυτή Οπωσδήποτε θα ήθελα να εκφράσω τη συγκίνησή μου για τον εργαζόμενο στη Μετάλ που αυτοκτόνησε πριν από λίγες μέρες με ένα συγκινητικό γράμμα που άφησε στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του. αυτή η χειρονομία, αυτό που έκανε, αυτό το τρομερό που συνέβη, μας αφορά όλους και με την γνωμοδότησή μας για το Χάλιβα, για τη Χαλιβουργία, ταυτόχρονα θα πρέπει να συλλογιστούμε και εκείνον και του συναδέλφους του. Και εκεί αναπτύσσεται μια ιδέα ότι υπάρχει μια υπερπαραγωγή, αλλά λοιπόν απαιτείται μια αναδιάρθρωση, αλλά υπάρχει μια αντίφαση η οποία εκφράζεται, γιατί σιγά σιγά να που διαλύονται εργαλεία εργασίας, αποδυναμώνονται και πρόθεσμα λένε ότι προσαρμόζονται στη συγκυρία, αλλά ως άλλη μεριά τι λέει, ότι θα έχουμε μια αύξηση 50% μέχρι το 2025 της ζήτησης χάλιβα. Άρα λοιπόν την αντίφαση αυτή θα πρέπει να την ξεπεράσουμε και μάλιστα όσο γίνεται πιο σωστά και να μην δεχτούμε έτσι τις δυνατότητες παραγωγής μας να τις καταστρέψουμε σαν κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να συμβεί και δυστυχώς ανέφερα ήδη ένα σλιβερό γεγονός αλλά υπάρχουν και πολλές χαλιβολίες που κλείνουν ε, χιλιάδες εργαζόμενοι χωρίς δουλειά, νέοι χωρίς μέλλον και χάνουμε και γνώση για το μέλλον επίσης αγορές ταυτόχρονα που τις κατακτούν ε, που προέρχονται από άλλες χώρες ή άλλες υπήρους. Τώρα οι πέντε προτάσεις ε, της γνωμοδότησης. Μέσω της πρώτης εκφράζεται μια ιδέα, τη γίνεται προσπάθεια τουλάχιστον, ότι όλοι μαζί, τα τρία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δράσουμε από κοινού συντονισμένα για όλα αυτά τα στοιχεία και όχι όπως κάνουμε μέχρι τώρα τμηματικά αυτό συνηθίζουμε ανάλογα με τις ε, γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμεί οι ίδιοι εδώ στο Κοινοβούλιο γιατί ασχολούνται διαφορετικές ε, επιτροπές με το θέμα αυτό. Το δεύτερο τμήμα έχει σχέση με αυτό που βλέπουμε από την λήξη της συνθήκης ΕΚΑΧ ε, που έλεγε ποιες ήταν δυνατότητες για τη βιομηχανία σήμερα. Δεν μπορεί κανείς πια να υποστηρίξει ανοιχτά δημόσια αυτό τον ε, τομέα που είναι όμως στρατηγικού χαρακτήρα και άλλοι ανταγωνιστικοί σήμερα τομείς, έτσι ε, τουλάχιστον θεωρούνται, αλλά αυτοί υποστηρίζονται από το δημόσιο, όπως η περίπτωση της αλουμίνας. Και θα πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα και εμείς ε, τι προτείνουμε να γνωμοδοτήσουμε με τη δυνατότητα επίσης στήριξης αυτού του στρατηγικού τομέα. Τρίτο θέμα επειδή δεν υπάρχει στήριξη, τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει ανάγκη να προσαρμοστεί κανείς στη συγκυρία με μια αναδιάρθρωση, ξέρουμε όμως τις συνέπειες. Και αρκετές φορές ε, δεν υπάρχουν προκαταρτικά ή στη συνέχεια συνοδευτικά μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστεί κανείς και πάλι την έκθεση του Αλεσάνδρου Σύρκας σχετικά με τις συνθήκε που επικρατούν ανάμεσα ε, για την ε, μεταβολή αυτή, την αλλαγή αυτή, την βιομηχανική. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων τι είπε ότι την έκθεση αυτή την υποστήριζε. Δυστυχώς όμως ε, δεν θα πρέπει έτσι να απαξιεί αυτό το κείμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να το λάβει υπόψη της και μάλιστα τάχιστα. Τέταρτο σημείο τώρα. Για, την, ε, ε, για τους εργαζόμενους και το πού θα εργαστούν τώρα θα πρέπει να, εμφαν, να υπάρξουν κονδύλια και με το Ταμείο αυτό προσαρμογής ε, στην παγκοσμιοποίηση δεν θα πρέπει να είναι μια κακή πολιτική, θα πρέπει, δεν θα πρέπει να μειωθεί το επίπεδο της στήριξης και το τελευταίο, αυτό που ζητάμε στην Επιτροπή μας εδώ και καιρό, με μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική που να αφορά την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες τις δυσκολίες, τη βαριά αυτή εργασία στη χαλιβουργία και πώς επηρεάζει η υγεία των εργαζομένων. Και υπάρχει και το στρες άλλωστε και η μειοσκελετική για τα προβλήματα και όλες αυτές οι συνέπειες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν υπολογίζει κανείς και το για το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Ε, αυτά θα πρέπει όλοι μας να τα δούμε και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε συμπληρωματικά και με τροπολογίες. Ευχαριστώ συνάδελφε. Επόμενο ο Φρίντριχ από τους ε, σοσιαλ, σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ. Καταρχήν, πριν να μπω στην ουσία του θέματος, ε, θα ήθελα να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο Και εγώ καθώς είμαι από έχω στενή επαφή με ναι, τα άτομα που εργάζονται στη χολιβουργία και με το γεγονός αυτό το τραγικό. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας επενθυμίσει ότι το κλείσιμο προκαλεί απελπισία στους εργαζόμενους ε, και θα πρέπει να αντιδράσει απέναντι στο κλείσιμο των ε, εργοστασίων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μπορούμε να λάβουμε μέτρα για να υπάρχει ψυχολογική βοήθεια που θα δίνεται σε αυτά τα άτομα. Σε ό,τι αφορά τώρα το σχέδιο γνωμοδότησης του συναδέλφου εδώ, θα ήθελα πάρα πολλά από αυτά τα θέματα που αναφέρονται εδώ να είναι θέματα με τα οποία ασχολείται δυναμικά η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχέδιο της γνωμοδότησης ε, έχουμε την διατύπωση ότι ε, είναι αφοπλισμένη κομισιόν έναντι στο φαινόμενο της ε, αναδιάρθρωση, δημιουργία βασικών κανόνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το θέμα της αναδιάρθρωσης αναφέρθηκε επίσης ότι πρέπει να υπάρχουν συνεχείς για την επαγγελματική κατάρτιση Τώρα εδώ βλέπω όλα αυτά τα θέματα και με θα υποστηρίξω και θα ενισχύσω τα σημεία αυτά. Και σε σχέση με την στρατηγική των πολυεθνικών, εμείς ε, βλέπουμε εδώ ότι αποφασίζουν περισσότερο να κλείσουν παρά να πουλήσουν ε, τα εργοστάσια. Αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην γνωμοδότηση και θα πρέπει η δημόσια αρχή να συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία για να μπορούμε να έχουμε χρόνο έτσι ώστε να βρεθούν νέοι ιδιωτικοί επενδυτές και να δοθεί νέα δυναμική σε μια εγκατάσταση. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί το φαινόμενο φαινόμενο του και Επίσης πρέπει να πούμε ότι αν η επένδυση στο τομέα έχει υψηλή προσθέμενη αξία, είναι θεμελιώδης και δεν πρέπει να μην αμελούμε τις επενδύσεις στο βασικό τομέα, στους βασικούς τομείς. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε την αναφορά στην έκθεση ΣΕΡΚΑΣ για τον κοινωνικό διάλογο και επίσης ε, και συμφωνώ και με την αναγκαιότητα να υπάρχει ψυχολογική παρακολούθηση των ατόμων αυτών και θα πρέπει να έχουμε μια πραγματική κοινή βιομηχανική πολιτική με τον κατάλληλο προπολογισμό, συντονισμό σε παιδό και την κατάλληλη νομοθεσία. Με τροπολογίε σε αυτά τα σημεία θα συμβάλλω και εγώ, αλλά ακολουθώ την ίδια φιλοσοφία με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ Φρεντερίκ. Ο κύριος Μπένιον, εξ των φιλελευθέρων. Um, Να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για τη γνωμοδότησή του για το τόσο σημαντικό αυτό θέμα. Νομίζω ότι η χαλιβουργία είναι και θα παραμείνει σημαντική στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντική και για άλλους τομείς όπως ε, για την μηχανουργία, κατασκευαστικό τομέα. Εξάλλου είναι σημαντική και για τις ανώσμες πηγές ενέργειας γιατί χρειαζόμαστε ισχυρή χαλιβουργία. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι υπήρξαν κάποιες δύσκολες ε, εποχές ε, και έλαβε υπόψη αυτά που λέει ο κύριος ε, σχετικά με τη στάση των ε, πολυεθνικών ε, στην περίπτωση του κλεισίματος ορισμένων βιομηχανιών. Είδα επίσης τι είπε και για το dumping, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα σε αρκετούς τομείς. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες σημαντικοί και δεν νομίζω ότι είναι σωστό να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα και μόνο παράγοντα. Η έκθεση εστιάζεται και στο ρόλο της διεύθυνση του management που προσπαθούν να προσποριστούν κέρδη εις βάρος ε, των ε, μισθών. Προφανές είναι αυτό, δεν πρέπει να σε εκπλήσει, οι manager πάντα κέρδη αναζητούν υπάρχει μια ε, ολόκληρη σειρά περίπλοκων ε, θεμάτων. Ε, ένα από τα προβλήματα είναι η προσφορά και ζήτηση, ίσως και το dumping και ίσως και οι τιμές της ενέργειας που διαφέρουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να τους εξετάσουμε αυτούς τους παράγοντες αντί να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα και μόνο. Επίσης είδα την ανακοίνωση της Επιτροπής επί του θέματος και διαπίστωσα ότι η Επιτροπή ήδη αναφέρεται στο ρόλο των κρατικών ενισχύσεων ε, σε σχέση με την ε, ανεργία και την ε, δημιουργία θέσεων εργασίας. Τέλος, συμφωνώ ότι τα κοινωτικά κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό την εποχή της βιομηχανικής μετάβασης. Γι' αυτό λοιπόν προσβλέπω στο να συνεργαστώ επί του θέματος μαζί με τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρω αν κάποιος... Ε, παρακαλώ, εσείς έχετε το λόγο. Στα γαλλικά θα μιλήσω. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας ε, για αυτή την απόφαση να συμμετάσχει και να εκφράσει αυτή την νομοδότηση Πελεγκρίνη σχετικά με τις πρώτες και τα μέταλλα υπεύθυνο και υποστηρίζω τα όσα είπε ο εισηγητής ε, σε μεγάλο μέρος και ένα σημείο στην αρχή συμφωνούμε για την ανάγκη ότι χρειάζεται μια συνολική αντιμετώπιση γιατί μερικές φορές είχαμε μονομένες πολιτικές και στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μερικές φορές τι γίνεται έχουμε γενικά αποτελέσματα αρκετά σημαντικά και αυτά στους διάφορους τομείς και στα τμήματα της ε, Επιτροπής Υπηρεσίες δεν πραγματοποιείται ο διάλογος που θα έπρεπε να πραγματοποιείται. Και αυτά μετά από το πρόγραμμα δράσης που έχετε μπροστά σας, να πούμε ότι ολοκληρώσαμε τη μελέτη επιπτώσεων σχετικά με διάφορες νομοθεσίες για το χάλιβα και τα έχουμε στο site web, site web της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δείχνουμε πώς επηρέασαν όλες οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες τα πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Για πρώτη φορά οι ενέργειες αυτές έγιναν από την Επιτροπή ο Χάλιβας που είπατε μερικές φορές τον είχαν παραμελήσει σαν τομέα και τώρα όμως μπήκε στην πρώτη γραμμή. Είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτή η μελέτη και που δείχνει ότι κυρίως σε περίοδο κρίσης επηρεάζεται αρκετά η Ευρωπαϊκή επηρεάζει αρκετά τα πράγματα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε αυτό. Τελευταίο αυτό που είπατε για τον τομέα μετά από την λήξη της ισχύω της συνθήκης ΕΚΑΧ. Ε, όπως το είπε ένα από τους βουλευτές σας, εντάξει, μπορούσε να δίνει κάποια βοήθεια στην έρευνη, και στην ανάπτυξη, ας πούμε, αλλά η Επιτροπή προσπαθεί να ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση για τη βοήθεια στην αναδιάρθρωση. Θα αποτελέσει ένα βήμα να δούμε αν θα πρέπει ο Χάλιβας και πάλι θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτόν τον τομέα να διάδοξει τη βοήθεια. Εντάξει και θα μπορεί κανείς για να εκφράσει την απόψή του. Ανάμεσα από τις έξι προτεραιότητες της δικές μας στο πρόγραμμα δράσης για το Χάλιβα, η κοινωνική διάσταση είναι απόλυτη προτεραιότητα. Αυτό το τραγικό γεγονός της Λιέγης πριν από λίγες μέρες η αυτοκτονία αυτή έδειξε ότι είναι κάτι το συγκεκριμένο αυτό το πρόβλημα και η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να προσχεθεί για δύο πρώτα θέματα. Πρώτα απ' όλα η αναδιάρθρωση που απαιτείται έτσι και αλλιώς ε, γενική, βαθιά ε, και δεύτερο γιατί όπως γνωρίζετε θα υπάρξει μία μετάβαση προς ε, ηλεκτρικές καμίνους και υπάρχουν αρκετοί τρόποι για την παραγωγή, αλλά αυτές οι ηλεκτρικές κάμινοι, δεν ε, ε, βέβαια χρησιμοποιούν λιγότερα εργατικά χέρια δυστυχώς γιατί πώς να το πούμε είναι labor intensive λιγότερο ε, και όχι μόνο αναδιάρθρωση αλλά η κοινωνική διάσταση είναι και η σχετική εκπαίδευση εκεί θα υπάρχει μια γνώση που θα πρέπει να διατηρηθεί στην Ευρώπη και θα πρέπει αυτό επαναλαμβάνω να διατηρηθεί. Τελευταίο σημείο τώρα που είναι ουσιαστικά δύο σημεία. Όπως ε, το είπαμε παρατηρείται μια κρίση τώρα υποφέρει ο χάλιβας γιατί όλοι οι τομείς που έχουν άγια από χάλιβα δηλαδή δομές, ε, τα αυτοκίνητα έχουν πρόβλημα λοιπόν και η ζήτηση χάλιβος μειώνεται αλλά όπως είπαμε στο πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής μέχρι το 2030 θα σημειωθεί ιδιαίτερα αύξηση της ζήτησης στον τομέα αυτό και θα πρέπει να είναι δική μας, το δική μας την αγορά θα πρέπει σαν δεύτερη παραγωγή εμείς στην Ευρώπη να διατηρήσουμε τη θέση αυτή. Και όπως το είπε ένας από τους βουλευτές, δεν πρέπει να έχουμε να κρατήσουμε μια προστατευτική πολιτική, θα πρέπει όμως να μπορέσουμε να μηνθούμε εμπορικά. Και το γνωρίζετε ότι πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια αλλαγή των μέσων προστασίας ε, του εμπορίου μας και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να υιοθετήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτά τα μέτρα. Αυτά λοιπόν και σε αυτά θα αρκεστώ. Ο εισηγητής Πατρίκ δύο λεπτά όμως πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία μετά. Γίνεται αυτό. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που κατέθεσαν την άποψή τους. Διαπιστώνω ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλες αποκλήσεις στις απόψεις μας. Έχουμε λοιπόν μια καλή βάση εργασίας. Άκουσα με προσοχή τα όλα όσα υπόθηκαν και κάποιες από τις προτάσεις που έκανε ο κ. Νταρντέν, κυρίως ό,τι αφορά τα διακυβεύματα της ε, κοινή βιομηχανικής πολιτικής, ό,τι αφορά το θέμα της εμπορικής πολιτικής Ίσως θα έπρεπε να ενισχύσουμε αυτή την πτυχή, γιατί η αγορά όπως έχει σήμερα μας θέτει σε μια κατάσταση ανταγωνισμού που δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε. Έτσι λοιπόν συμφωνώ να υιοθετήσω όσα υπόθηκαν για το θέμα αυτό και τις επόμενες εβδομάδες θα εργαστούμε από κοινού για τη βελτίωση αυτής της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ η διορία για την κατάθεση τροπολογιών 24 Οκτωβρίου στις 12 το πρωί. Τώρα περνάμε στην ε, ψηφοφορία. Το σημαντικότερο από όλα είναι βέβαια να έχετε τις κάρτες σας. Φαντάζομαι ότι όλοι τις έχετε. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει το θέμα της ε, κοινωνικής διάστασης, ε, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Είναι η έκθεση της συναδέλφου Περές της ε, Προέδρου μας ε, και έρχομαι στον πρώτο από τους ε, δύο καταλόγους που έχουμε. Ελπίζω να έχετε όλοι μπροστά σας τον ίδιο κατάλογο. Πρόκειται για το θέμα υπαρθμών 1 και υπαρθμών 7. Προτείνουμε να ψηφιστούν unblock. Ποιος είναι υπέρ, κατά, μισό λεπτό, καλύτερα ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πολύ ωραία. Το αποτέλεσμα παρακαλώ. 17 ναι, 12 όχι, 12 κατά. Τώρα, οι δύο της κυρίας Κορνέλισεν και άλλων υπέρ, κατά και εδώ πάλι ε, ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. ψηφίζει. Έκλεισε η ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα παρακαλώ. Απορρίπτεται. Το 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν αποχές. Η 4 αποσύρθηκε. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Η 5. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 6 αποσύρθηκε. Η 8 είναι συμβατή. Ε, υπέρ ε, καλύτερα ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε για την 8 παρακαλώ. Η έξι αποσύρεται, είπατε. Πότε το είπατε. Ε, ψηφίζουμε για την Οκτώ. On the Commission communication. Uh, we've got them in the wrong order, that's why. Ah, that's why. Good. Okay, so just now. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την Οκτώ του Φιλ Μπένιον. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα παρακαλώ. 18 υπέρ, 16 ε, κατά. Η 9 αποσύρθηκε. Η 10 κορνέλησαν και άλλων. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Λοιπόν, καλύτερα ε, να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε. Το αποτέλεσμα παρακαλώ. 17 ναι, 16 κατά. Ε, ψηφίστηκε, υπερψηφίστηκε με μία ψήφο διαφορά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τώρα για το σύνολο της έκθεσης. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πολύ ωραία. Έκλεισε Ψηφίστηκε. Πάει αυτό. υπερψηφίστηκε. Πάμε τώρα στην δεύτερη έκθεση. Μπέρες και μετά θα ξεκινήσουμε unblock για την 1 και τη 10 υπέρ παρακαλώ κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίζουμε Ψηφίζουμε για την 1 και την 10 παρακαλώ. Υπερψηφίστηκε. Πάμε στην υπαρτιμόν 2. Μαρή Κορνέλησιν και άλλοι. Υπέρ παρακαλώ. Το αποτέλεσμα παρακαλώ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφορίας. 17 ναι, 16 κατά και 2 αποχές. Εγκρίθηκε. Οι δύο, Κορνέλισεν και άλλοι. Υπέρ παρακαλώ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Abstimmung geschlossen. Έκλεισε ψηφορία. Und das Ergebnis heißt 18 Ja und 17 Nein und eine Enthaltung. Auch hier akzeptiert. Εγκρίνεται. Η τρία. Σαμπαέρι, υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστούμε κατά ηλεκτρονικά. So, bitte schön, Abstimmung ist eröffnet. Und die ist geschlossen. Und das Ergebnis? Το αποτέλεσμα παρακαλώ. 17 ja, 20. Απορρίπτεται. Πάμε στην υπαριθμό 5, Εμερ Αποσύρθηκε 4, Σαμπαέρι, υπέρ, κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Το 7. Ο ίδιος ε, εισηγητής, ο συντάκτης της τροπολογίας, ο κ. Σάμπα Έρη, Απορρίπτεται. Η 6. Φιλ Μπένιον. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Σαμπαέρι 8. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 9 αποσύρθηκε. Η 11 Υπέρ της 11 παρακαλώ. Απορρίπτεται. Η 12 αποσύρθηκε. Η 13 Φιλμπένιον υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 14 κατά. Δεκατέσσερα παρακαλώ. Δεκαπέντε υπέρ, είκοσι κατά και οι δεκαπέντε υπέρ κατά απορρίπτεται. Περνάμε στην τελική ψηφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφορία. Το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην προφορική ερώτηση ε, ισπανικά θα μιλήσετε, γι' αυτό μισό λεπτό να βάλω και εγώ τα ακουστικά μου. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν ε, ξέρετε τι ακριβώς κάνουμε, δηλαδή θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα ψήφισμα ε, για να διαφοροποιηθούμε. Όμως τώρα δεν ε, ξέρω αν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια διαδικασία και το επιδυναμώναμε καμία πολιτική διαδικασία. Δηλαδή τώρα όταν έχουμε μια ψηφοφορία τόσο στενή, ουσιαστικά είναι το ίδιο σαν να εγκρίνουμε μια τροπολογία κατά ενός κειμένου, δηλαδή χρειάζεται η ίδια πλειοψηφία μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαμπαόρη. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ψηφίσαμε. Άρα λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας το αποτέλεσμα. Και δεν είναι τυχαίο ότι καταψηφίσαμε αυτό γιατί πολλά στοιχεία ε, είναι κατά αυτών των ε, βασικών αρμοδιοτήτων των κρατών μελών ε, και ε, να μην ανακατευθούμε σε αυτό και στην, σε εκλογέ των σοσιαλιστών στην εκστρατεία τους. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η δεύτερη παρατήρηση είναι γελία και η πρώτη είναι εννοητή. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ζητάνε από το Συμβούλιο. Αν δεν μπορούμε να ζητήσουμε από το Συμβούλιο ποια είναι η άποψή του σε μια ανακοίνωση πάνω τη Επιτροπή, ε, τότε σύμφωνα με αυτό που λέει ο Συνάλφος θα έπρεπε να το κλείσουμε εδώ, να το βουλώσουμε και είναι εντελώ διαφορετικό το πρότυπο από ότι αυτό εδώ. Διαφορετικά δεν έχουμε καμία άποψη δηλαδή εμείς να εκφράσουμε, έτσι. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε για το επόμενο θέμα. Είναι προφορική η τροπολογία. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν. Ακούσαμε λοιπόν την πολιτική ανταλλαγή απόψεων και πάμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης. Αν συμφωνείτε, η έκθεση Τατιάνα Στανόκα ε, σχετικά με τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνα εργατικού δυναμικού στην κοινότητα. Η τέσσερα υπέρ Τατιάνα Στανόκα. Κατά. Πολύ ωραία, σαφής η πλειοψηφία, απορρίπτεται. Πάμε τώρα στα σημεία 5 μέχρι 8. Ψηφίζουμε και για όλα αυτά τα σημεία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται με σαφήνεια. Πάμε τώρα στην προφορική τροπολογία για τον προϋπολογισμό υπαριθμών 2. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο πρόβλημα επ' αυτού. Από βλέπω όχι. Ε, για τον προϋπολογισμό υπαριθμών 2. Υπέρ παρακαλώ σαφής η πλειοψηφία, αποδεκτό. Πάμε τώρα στην συμβαστική ε, υπέρ παρακαλώ, σαφής η πλειοψηφία. Πάμε στην F, η συμβαστική F, σαφής η πλειοψηφία. Η G, όπως Gustav, και εδώ σαφής η πλειοψηφία. Στην 24 πάμε, στην κυρία κυρία Σάρη, υπέρ παρακαλώ, σαφής η πλειοψηφία. Πάμε στην υπαριθμόν συμβαστική Α, σαφής η πλειοψηφία, στην Β και εδώ σαφές το αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στην υπαριθμόν 2 της εισηγήτριας, υπέρ παρακαλώ. Κατά απορρίπτεται. Πάμε στην συμβαστική σε υπέρ παρακαλώ. Σαφής η πλειοψηφία. Η δέλτα και αυτή είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ε, δεκτό, έχουμε τη 18, Κοστέλο, υπέρ παρακαλώ, σαφής η πλειοψηφία. Και πάμε τώρα στη συνολική, στην ψηφορία του συνολικού ψηφίσματος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Για το σχέδιο της έκθεσης ε, έκλεισε η ψηφοφορία. 22, μισό λεπτό, 32 υπέρ, 2 κατά, 3 αποχές και το ίδιο ισχύει για το ε, ε, νομισματικό ψήφισμα. Ψήφισμα έκλεισε η ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα παρακαλώ. 30 ναι, 2 όχι και 3 αποχές. Και πάμε τώρα στο κατά πόσον θέλουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις ή όχι. Ε, τουλάχιστον 26 πρέπει να είναι παρόντες, σαφές, ε, ψηφίζουμε. Έκλεισε η οχι τουλαχιστον 26 πρεπει να ειναι παροντες σαφες ψηφιζουμε εκλεισε η ψηφοφορια 31 υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές και συγχαρητήρια σε όλους τους εισηγητές. Τώρα, το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης είναι η έκθεση Jean Lambert. Δεν είναι εδώ ο Jean, αλλά η έκθεση είναι εδώ. Πάμε στη συμβαστική Β, ε, υπέρ παρακαλώ. Ωραία. Εγκρίνεται η ΣΕ, υπέρ, κατά, Σαφές το αποτέλεσμα. Υπέρ. Πάμε τώρα. Ε, πάμε στην 14. Ε, Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Σαφές το αποτέλεσμα. Υπέρ. 15 της Γιούτα. Υπέρ παρακαλώ κατά η 16 υπέρ κατά σαφές το αποτέλεσμα συμβιβαστική δέλτα υπέρ παρακαλώ σαφές το αποτέλεσμα υπέρ η 18 Σαμπασόγκορ υπέρ κατά μισό λεπτό περισσότερη κατά Σάμπα. 20. Φιλ Μπένιον. Υπέρ. Κατά. Σαφές το αποτέλεσμα. Υπέρ. Και της κυρίας Αντιγόνης. Υπέρ. Κατά. Υπέρ. Πάμε στην ε. 25 ε, της εισηγήτριας. Μισό λεπτό, λέει ο πρόεδρος. Όχι, μισό λεπτό. Δεν ψηφίζουμε, αλλά κανονικά θα ψήφιζαν όλοι υπέρ, λέει ο πρόεδρος. Πάμε στη συμβαστική F. Ε, σαφές το αποτέλεσμα, υπέρ, η 1 της Jean Lambert, ε, υπέρ, σαφές το αποτέλεσμα, υπέρ και συμβιβαστική α. Και εδώ ε, σαφές το αποτέλεσμα υπέρ και οι τρία της ε, Αντιγόνης υπέρ κατά ε, υπέρ. Πάμε στο τελικό αποτέλεσμα της ε, Jean Lambert. Έκλεισε η ψηφοφορία. Λοιπόν, 33 υπέρ, 2 κατά. Συγχαρητήρια στην Τζιν Λαμπερτ. Μπορείτε να τις διαβιβάσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στην έκθεση Κάζα. Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Ελληνικό Εμπόλιο προς όφελος όλων των παραγόντων. Και ξεκινάμε με τη συμβαστική α. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Η υπαριθμόν 3. Μίλαν καπτσνοχ, υπέρ. Κατά. Νομίζω περισσότερο περισσότεροι υπέρ. Καλύτερα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Ψηφίζουμε, Αλεσάνδρο. Θέλω απλά εσείς να διευκρινίσετε ποιος είναι ο αριθμός της συμβαστικής πρότασης. Το 3 λέει ο πρόεδρος. Το 3. Ψηφίζουμε για το 3. Ε, γι' αυτό είναι καλό να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 3. Έκλειση ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα παρακαλώ. 20 ναι, 16 κατά, καμία αποχή. Πάμε στην τροπολογία του αδέλφου Πουπάκη, η 4 υπέρ παρακαλώ, κατά, μάλλον ήταν σαφές αποτέλεσμα, όλοι υπέρ. Η 5 ψηφίζουμε σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, σαφές το αποτέλεσμα, υπέρ, για το δεύτερο τμήμα, υπέρ παρακαλώ, κατά, Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το 2. Έκλειση ψηφοφορία. 19 υπέρ, 17 κατά, καμία εποχή. Πάμε τώρα στη συμβαστική Β πολλών πολιτικών ομάδων. Υπέρ παρακαλώ, σαφές το αποτέλεσμα. Και η τροπολογία υπέρ του κυρίου Πουπάκη, υπέρ. Και εδώ σαφές το αποτέλεσμα η τροπολογία υπαριθμών 11 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ε, Κοτσολίνο, Ανδρέα, εισηγήτρια, υπέρ, σαφές το αποτέλεσμα, υπέρ. Και για το δεύτερο τμήμα, μισό λεπτό, με προφορική τροπολογία από τους ε, φιλελεύθερους. Ε, δεν διαφωνεί κανείς, άρα ποιος είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος με την προφορική τροπολογία, σαφές το αποτέλεσμα, υπέρ. Και το δεύτερο τμήμα λέει συστήνει να είναι σημαντική κοινωνική εταίρη. Υπέρ αυτού παρακαλώ. Μισό λεπτό. Κατά. Οι περισσότεροι είναι κατά, λέει ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, εμένα στο δεύτερο τμήμα, το πρώτο τμήμα εγκρίθηκε, πάει αυτό. Ο κύριος Σαμπαερή έχει να ρωτήσει κάτι επ' αυτού. Κοίταξτε, δεν ήταν απόλυτα σαφές. Το δεύτερο τμήμα λέει μαζί με την ε, προφορική τροπολογία. Άρα δεν χρειάζεται εδώ να ξαναψηφίσουμε. Ήδη ψηφίσαμε επ' αυτού. Νομίζω λοιπόν ότι για το δεύτερο τμήμα ήδη ψηφίσαμε και υπερψηφίσαμε. Ε, νομίζω έχει ήδη εγκριθεί. Απλά επειδή δημιουργείται κάποια σύγχυση στον κατάλογο, Λοιπόν, ψηφίζουμε για το ε, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφορία. 17 υπέρ, 16 κατά και 2 απόχέ. Και το δεύτερο τμήμα καλεί τα κράτη-μέλη, ε, όλοι υπέρ, εγκρίνεται. Πάμε στην 13, Έμα Κοστέλο, υπέρ παρακαλώ σαφές το αποτέλεσμα υπέρ η 14 και εδώ πάλι ε, προφορική τροπολογία από το συντάκτη υπέρ παρακαλώ. Πολύ ωραία. Σαφές το αποτέλεσμα υπέρ. Πάμε στη 15. Ε, υπέρ παρακαλώ, σαφές το αποτέλεσμα υπέρ, η συμβαστική C. Ευχαριστώ, ε, δεκτό. Η 20, πάμε στην 20, υπέρ παρακαλώ σαφές υπέρ 21 εδώ πάλι σε τμήματα για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά λίγη κατά αποδεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος του δευτέρου τμήματος έκλειση ψηφοφορία το αποτέλεσμα παρακαλώ 16 υπέρ, 15 κατά. Πάμε στη συμβαστική δέλτα υπέρ. Και τώρα πάμε στην 24. Είχα σκεφτεί να τα ψηφίσουμε όλα μαζί, αλλά δεν γίνεται. Ξεκινάμε την 24. Υπέρ. Σαφές το αποτέλεσμα. Υπέρ. 25. Υπέρ κατά. Υπέρ όλοι. 26 ή να ρωτήσω από την 26 να τα ψηφίσουμε όλα μαζί μέχρι το 31 τι λέτε όχι την 27 όχι εντάξει λοιπόν ας τα ξανακάνουμε όπως πρέπει 26 υπέρ σαφές το αποτέλεσμα υπέρ 27 υπέρ σαφές το αποτέλεσμα υπέρ 28 Κατά. Καλύτερα ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίζουμε για την 28. Έκλεισε ψηφοφορία. 23 υπέρ, 13 κατά, 29 παρακαλώ, υπέρ, κατά, καλύτερα ηλεκτρονική επαλήθευση για την 29 παρακαλώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση και έκλειση ψηφοφορία. 19 υπέρ, 13 κατά και 3 δήλωσαν αποχή. Η 30 τώρα παρακαλώ. Η 31 υπέρ σαφές και έχουμε ηλεκτρονική ψηφορία για το σύνολο του ψηφίσματος. Ψηφίζουμε παρακαλώ και έκλεισε ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα 34 υπέρ, 2 κατά και καμία αποχή. Και ε, έτσι ευχαριστούμε θερμά ε, τον Ντάβιτ Κάζα και ε, καλή ανάρρωση λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ich darf darauf hinweisen, die etwas später kamen, Θέλω να σας ε, επισημάνω ότι για αυτούς που ήρθατε αργότερα δεν θα ψηφίσουμε για την έκθεση Χάρκιν. Υπήρχαν κάποια προβλήματα, γι' αυτό και δεν υπάρχει στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, όσοι πρέπει τώρα ε, πρέπει να πάνε σε άλλες επιτροπές. Τελείωσαν οι ψηφοφορίες και θα συζητήσουμε τώρα για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Καταρχήν ε, θα έπρεπε να συζητήσουμε για την έκθεση την υπαρθμών 12, αλλά θα την ε, μεταθέσουμε λιγάκι, για λιγάκι αργότερα. Πάμε στην 20 και την 21 που όπως σας είπα προτάχθηκαν, το είχα πει προηγουμένως για όσους δεν είχαν έρθει ακόμα. Ο κύριος Νταρντάν έχει το λόγο. Έχεις δύο εκθέσεις, ε, Φιλίπ, ε, και περιμένουμε με αγωνία τις απόψεις σου. Φιλίπ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τις δύο να τις κάνουμε μία. για τις τροπολογίες πώς τις λαμβάνονται υπόψη αλλά να σας πω ποια είναι η γενική φιλοσοφία του σχεδίου γνωμοδοτησής μου τη γενική αυτή στρατηγική που στη σύνταξη και τις συμπληματικές τροπολογίες και στην ομάδα αυτές οι προτάσεις ε, δεν χρειάζονται να μπήσω γιατί περισσότερο άνοιγμα κλπ. Ε, οι εμπόδια δεν θα βελτιώσουν ε, την πρόσβαση στο χώρο αυτό και τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα σε σχέση τουλάχιστον με άλλους τρόπους μετάφορες και δεν θα μειώσουν το κόστος για τους χρήστες. Γι' αυτό λοιπόν στα πλαίσια αυτά εμείς ε, θα είχαμε να κάνουμε μια επιλογή. Είτε απλά και μόνο την απόψή μας να καθέσουμε για απόρριψη του σχεδίου, είτε μια άποψη, με διάφορες αποχρώσεις ε, και κάπως να αφαιρέσουμε ορισμένες προτάσεις ε, και νοήματα. Αυτό διαλέξαμε με τις βασικές ε, τροπολογίες και τις νοηματικές για να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε, πώς να επηρεάσουμε δηλαδή το τελικό οριστικό κείμενο. για τη διαχείριση την όλη. Ο στόχος μας ποιος είναι αυτό το συνικό τείχος ε, μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών και του διαχωρισμού τους και του αυτό πώς θα τα ξεχωρίσουμε και επίση τις υποχρεώσεις της δημόσιας ε, των δύο υπηρεσιών θέλουμε τρεις φάσεις. Πρώτα απ' όλα να δούμε την κατάργηση, την πλήρη των προτάσεων της Επιτροπής και οι εθνικές αρχές να μπορούν να αναθέτουν τα συμβόλαια και αν δεν είναι δυνατό δεύτερο επίπεδο με αύξηση του σωροφής και τρίτο και να αναβληθεί τρίτη φάση η προθεσμία να πάει αργότερα και υπάρχει μια προστασία έτσι και για το προσωπικό και την αλλαγή προσωπικού αλλού σύμφωνα με το δίκαιο αν υπάρχει κάπου αλλού κάποιος που να αναλάβει αυτήν την αγορά ενίσχυση κοινωνικού διαλόγου και με μια πιστοποίηση του προσωπικού και επίσης ε, αμοιβαία αντιμετώπιση, όλα αυτά ορισμένα παραδείγματα. Όσο με τις τροπολογίες που είναι και πολλές μάλιστα τη διαπιστώνω. Λοιπόν, για τη διαχείριση αυτή και για την υποχρέωση δημόσιας ε, υπηρεσίας ε, υπάρχει μια καλή σύγκληση με τις τροπολογίες του ΕΛΚ για τα κοινωνικά σύγκληση με τους πράσινους και την αριστερά και σχετικά με τους φιλελεύθερους ε, από εκεί κάπως περίμενα πώς το πω τώρα μετά από όσα άκουσα από τον συνάδελφο μετά από την παρουσίαση νομοδότησης ε, εκεί υπάρχουν αποκλήσεις και μάλιστα ριζικά αντίθετες απόψεις μερικές φορές ε, αυτό θα να πω και μάλιστα περιληπτικά τώρα. Εμείς προετοιμάζουμε συμβαστικά κείμενα για να δούμε με αυτές τις τροπολογίες πώς θα έχουμε θέσεις που θα συγκλίνουν περισσότερο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, περνάμε στον ε, κατάλογο των ομιλητών. Ο Ζως Μπάχ από το Λουξεμβούργο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Τόμας. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε μόλις τώρα στην Αλφος Φεντερίκ Νομίζω ότι βεβαίως και πρέπει να κάνουμε αυτήν την επιλογή. Εκείνος την έκανε την επιλογή. Εμείς ε, συμφωνήσαμε ε, και νομίζω μια πλήρης ε, απόρριψη σε αυτό το τόσο δύσκολο θέμα θα σήμαινε ότι δεν προχωράμε περισσότερο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι κατά τα επόμενα ετή πρέπει να βελτιώσουμε τους σιδηρόδρομους ε, στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Ο Φρεντερικ μίλησε για, τον, ε, για το κινέζικο τείχος και Γι' αυτό τον λόγο και εγώ στην Επιτροπή Μεταφορών λέω ότι δεν μπορούμε στην Ευρώπη να εισάγουμε ένα ενιαίο σύστημα σιδηροδρόμων. Υπάρχει μια ε, πληθώρα ε, δομών, ε, πολιτισμών και διαφόρων περιφερειακών ιδιομορφιών τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει και στα κράτη-μέλη να προσφέρουμε μια κάποια ευελιξία έτσι ώστε τα συστήματά τους να τα διαμορφώσουν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και για τους πελάτες και για τους εργαζόμενους. Γιατί αν δεν το κάνουν αυτό θα συνεπάγεται το επιπρόσθετο διοικητικό κόστος και δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Όσον αφορά αυτά που μας είπε ο κύριος Φρεντερίκ Νταρντά, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο στην περαιτέρω κατάρτιση του προσωπικού, στην πιστοποίησή του και να καταστήσουμε σαφές ότι όλα αυτά συνδέονται άμεσα και με τις συνθήκες εργασίας. Κατόπιν τούτου πρέπει να αναλάβουμε περισσότερες προσπάθειες. Σε περίπτωση εξαγοράς όλα αυτά είναι σημαντικά που σας είπα. Βεβαίως ε, εμείς στην Επιτροπή Μεταφορών επιμένουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει, να συνεχίσει να υπάρχει η απευθείας ανάθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει αν κρυθεί απαραίτητο θα πρέπει να υπάρχει μια περαιτέρω προστασία πέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει στην ε, κείμενη νομοθεσία. Εγώ σας λέω νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα και είμαι αισιόδοξο. Ε, θεωρώ ότι ο κύριος Νταρντά ε, θα καταθέσει από εκείνο με εμάς τροπολογίες προς όφελος των απασχολουμένων. Ε, αυτά εκ μέρους του ΕΛΚ. Τώρα, εκ μέρους των Θρηλευτέρων, παρακαλώ. Ο κύριος Ντεμπάκερ είναι σκιώδης για αυτούς τους δύο φακέλους αλλά είναι στο Τάλιν ε, για τις διαπραγματεύσεις για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών καθώς συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταφορών ε, και να πω ότι και εγώ και ο κύριος Μπέκερ ε, συμφωνούμε μάλλον έχουμε κοινέ αρμοδιότητες για το φάκελο αυτό στην αρμόδια Επιτροπή, την Επιτροπή Μεταφορών. Έχουμε λοιπόν καταθέσει πολλέ τροπολογίε για το άνοιγμα των αγορών, γιατί πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να ζήσει η αγορά το πλήρε δυναμικό τη. Εδώ αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι αλλαγή του μοντέλου. Επομένω, εργαζόμαστε σε μία βάση ε, που βασίζεται στις αποδείξεις ε, και αυτό έχει κατευθύνει τη θέση μας. Ε, ο Φιλίπ θέλει να τονίσει ότι το άνοιγμα των αγορών δεν οδηγεί στο κοινωνικό ντάμπινγκ, δεν το έχει κάνει. Αν δούμε και τα στοιχεία από Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι δύο χώρες που έχουν απελευθερώσει την αγορά τους, θα δούμε ότι σε αυτές τις δύο χώρες μόνο ε, ουσιαστικά μεγενθήθηκε η αγορά των σιδηροδρόμων και είναι ένα καλό παράδειγμα να δούμε. Οι χώρες αυτές ε, δεν ε, είχαν μια αδύναμη αγορά εργασίας, αλλά αυξήθηκαν οι δυνατότητες ε, και οι μισθοί και η θέσει εργασία, το επίπεδο απασχόληση, η σημερινή αγορά σιδηροδρόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί καλά και το να υπερασπίσουμε το status quo δεν θα βοηθήσει καθόλου την αγορά. Πρόκειται για ένα βαλκανοποιημένο σύστημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο χώρο σιδηροδρόμων, η χρήση των σιδηροδρόμων και τα δικαιώματα των επιβατών πρέπει να βελτιωθούν. Σήμερα ε, δεν ε, θεωρείται η ικανοποίηση των επιβατών ως πρώτη προτεραιότητα. Έτσι λοιπόν ε, τα δικαιώματα ανοιχτή πρόσβαση θα πρέπει να είναι ο κανόνα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν και δημόσιας υπηρεσίας. υπηρεσία. Το έχουμε κάνει αυτό στο Ρωμένο Βασίλειο και για τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και ήταν με μεγάλη επιτυχία. Είδαμε ω αποτέλεσμα να αυξάνεται η συχνότητα των υπηρεσιών. Όμως, είναι ε, θα πρέπει να, υπάρχουν, να υπάρχει και δυνατότητα και άμεσων αναθέσεων, αλλά θα πρέπει να γίνεται υπό συγκεκριμένε προποθέσει και θα καταθέσουμε τροπολογίε προ αυτό. Θα πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα τη Κομισιόν, γιατί αν έχουμε περαιτέρω καθυστερήσει, θα αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα στην αγορά των σιδηροδρόμων. Ο Φιλίπ επίση καταθέσει μια τροπολογία για να εισαγάγει ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσία ε, όταν ε, υπάρχει απεργία και θα υπάρχει τότε εγγύηση για τους επιβάτες όταν ταξιδεύουμε με το τρένο. Υπάρχουν κάποιοι ευρωπαϊκοί κανόνες για το προσωπικό και το τέταρτο πακέτο αφήνει τους κανόνες ως έχει. Αυτό αποτελεί συνδυασμό με τους εθνικούς κανόνες και τα κοινωνικά πρότυπα και ουσιαστικά δεν ε, χρειάζεται περαιτέρω ρυθμίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, ε, μόνο αν υπάρχει συνεργασία μεταξύ του ε, διευθυντή και των ε, επενδυτών θα υπάρχει καλύτερη βελτίωση. Σε ό,τι αφορά το τεστ της ηρωπίας, εγώ έχω ε, συνυπογράψει τροπολογίες για να έχουμε και το startup μιας δημόσιας υπηρεσίας. Θέλουμε επίσης και οι υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης να λάβουν την απαραίτητη στήριξη. Και φυσικά ο Φιλίπ θα συζητήσει αυτές ε, τις τροπολογίες με τον συγητή εκ μέρου των Πρασίνων, η η κυρία Σρόιντερ. Λοιπόν, εγώ έχω καταθέσει μια ολόκληρη σειρά τροπολογιών και θα ήθελα ο εισηγητή ε, να μου πει ποια είναι η γνώμη του ε, όσον αφορά αυτές τις ε, τροπολογίες. Αυτό για μας, για την πολιτική μας ομάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι δικές μου οι τροπολογίες αφορούν στο θέμα του διαχωρισμού ανάμεσα στην υποδομή και στον πάροχο στους ε, παρόχους ε, των σιδηροδομικών υπηρεσιών. Εμείς λοιπόν στηριζόμαστε στο εξής, στο ερώτημα τελικά τι γίνεται με τους εργαζόμενους. Νομίζω ότι είναι σαφές, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο πακέτο το οποίο έχει πάρα πολλές επιπτώσεις στα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Πράγματι υπάρχει αυτή η τάση του εξευρωπαϊσμού, άρα δηλαδή και σε αυτό τον τομέα θα πρέπει να υπάρχουν ε, κατώτατα όρια και κατώτατες ε, προϋποθέσεις απασχόλησης. Σε σχέση με αυτά που είπατε για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση, συμφωνώ και εγώ, αλλά επίσης ε, και για το ότι θα πρέπει να προσφέρετε προστασία στους οργαζόμενους οποτεδήποτε προκύπτουν διαρθρωτικές αλλαγές η τεχνογνωσία των εργαζομένων δεν μπορεί να πετιέται στα σκουπίδια. Το λέω αυτό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ειδικού και η διασύνδεση πολλών πραγμάτων όπως ε, παραδείγματο χάνει η διασύνδεση ε, των συνεργείων με τις μονάδες των παρόχων, αυτά είναι άμεσα συνδεμένα μεταξύ τους και αν τα χωρίσουμε θα υπάρξει μειονέκτημα, μεγάλο μειονέκτημα. Δεν ξέρω αν θα ε, ξακολουθεί να υπάρχει απαραίτητη τεχνογνωσία και αν όχι ε, θα είναι μεγάλη απώλεια αυτό για την Ευρώπη. Θέλω λοιπόν να γνωρίζω την άποψη του εισηγητή επ' αυτού. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, αυτό έρχεται σε λάθος στιγμή, είναι περιττό. Έχουμε ένα άνοιγμα των αστικών μεταφορών στην Ευρώπη. Παλαιότερα ως κοινοβούλιο είπαμε ότι δεν μπορεί να είναι όλα ανοιχτά ε, γιατί εμείς ε, έχουμε την υποχρέωση κυρίως ε, για μελετού περιοχές να διατηρηθούν κάποιες ε, συνδέσεις, διασυνδέσεις. Εντάξει, μπορεί αφορά απαραίτητα το Λουξεμβούργο, αλλά άλλες περιοχές ε, που έχουν μικρά, μικρά χωριά, απομακρυσμένες περιοχές και άνθρωποι το θέλουν και αυτοί το βράδυ ή δυνατόν να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Εμείς λοιπόν ως Κοινοβούλιο όταν ήρθε το πρώτο άνοιγμα είπαμε ότι για αυτές τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές ε, έχουμε δεσμευτεί να τους διατηρήσουμε εκεί τους ανθρώπους αυτούς. Αυτές οι περιοχές ε, εξαρτώνται ιδιαίτερα από μας Ας πούμε, έχω κατά νου κάποιες ε, περιοχές στις Άλπεις που αυτά τα μέρη δεν θέλουν να αποκοπούν. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο βρήκαμε μια ειδική ρύθμιση, την οποία ρύθμιση η Κομισιόν τώρα πέταξε, την αγνόησε. Εγώ αυτό το θεωρώ πρόβλημα. Γι' αυτό κατέθεσα ε, τροπολογίες που υπογραμμίζουν αυτή την υποχρέωσή μας ε, διατήρησης αυτών των ανθρώπων. Στην Ευρώπη Λένε μερικοί ότι θα πρέπει να μπορεί κανείς να ταξιδέψει από το ένα ε, σημείο στο άλλο της ε, Ευρώπης με ένα και μόνο εισιτήριο. Εγώ το στηρίζω αυτό. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ε, αν θέλουμε να διασυνδέσουμε δύο περιοχές για να μπορεί κανείς να πάει από τη μία περιοχή στην άλλη, αυτό ήδη και μόνο αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Πολλές φορές ε, οι τιμές ε, στα μεγάλα αστικά κέντρα ε, είναι πολύ ψηλότερες από αυτές που μπορούν να καταβάλουν άτομοι της επαρχίας και πολλοί άνθρωποι εξαρτώνται τέλος πάντων από αυτές τις μεταφορές. Υπάρχει το κοινωνικό στοιχείο, το κοινωνικό, η κοινωνική διάσταση όπου αν κάποιος δεν ανήκει στα πλούσια στρώματα ε, θέλει να χρησιμοποιεί τα δημόσια μέσα μεταφοράς γιατί μέχρι εκεί μπορεί να πληρώσει. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε αυτές οι απομακρυσμένες περιοχές να έχουν ε, βασική διασύνδεση όχι μια φορά τη βδομάδα, το πρωί και το βράδυ να μπορούν και οι άνθρωποι το βράδυ να πάνε στο θέατρο και πολλά άλλα. Κατά την άποψή μου αυτά είναι καθοριστική σημασία. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σας είπα κατέθεσα τροπολογίες και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το τι θα γίνει γιατί αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι να διατηρηθούν κάποιες υποδομές που θα εξυπηρετούν τους ανθρώπους και για όλους αυτούς τους λόγους με ενδιαφέρει να ξέρω ποια είναι η άποψη του εισηγητή. Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ίσως μπορείτε να μας πείτε και το όνομά σας για να το καταγράψουμε στα ε, πρακτικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. κύριε Πρόεδρε. Τον εισηγητή τον ευχαριστώ για την εργασία του επί των δύο προτάσεων αυτών, όπως και τα μέλη της Επιτροπής σας που υπέβαλαν τροπολογίες. Είναι πολύ σημαντικά κείμενα για το αστυνομικό τομέα, γιατί έχουν να κάνουν και με την όλη δομή των οργανισμών σιδηροδρόμων και με την όλη δομή και τη λειτουργία βέβαια της αγοράς και των υπηρεσιών των περιφερειακών. Πριν να κάνω εσμένα σχόλια για αυτά τι σημαντικές τροπολογίες, να πω ξεκινώντας κάτι για ένα θέμα το κοινωνικό σε αυτές τις προτάσεις. Οι στόχοι των προτάσεων της Επιτροπής ποιοι είναι να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες της ε, δρομικών ε, συνδέσεων και να την προσφέρουμε αυτή τη βελτίωση στους πολίτες. Όλα αυτά βέβαια σεβόμενοι απόλυτα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Να υπενθυμίσω κάτι ότι η νομοθεσία ευρωπαϊκή προβλέπει ήδη ρυθμίσεις προστατεύουν ε, τους εργαζόμενους για το 1372-2007 αυτόν τον κανονισμό για μια αλλαγή της απασχόλησης των εργαζομένων από τη στιγμή που θα αλλάξει ο φορέας. Άρα λοιπόν προστατεύεται ε, ο εργαζόμενος σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν πολλές διάφορες ρυθμίσεις προστατεύουν τους εργαζόμενους και σε εθνικό επίσης επίπεδο ειδικότερα δε στα πλαίσια ορισμένων συλλογικών συμβάσεων των συλλογικών συμβάσεων κάτι να τονίσω τα κράτη-μέλη που έχουν ανοιχτό ανταγωνισμό στην αγορά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και Σουηδία κυρίως ε, δεν ε, χάσαμε θέσεις εργασίας. Αντίθετα, απασχολούνται περισσότεροι στον τομέα αυτό το συνδρομών, όπως πολύ σωστά ο κ. Πενιών το υπενθύμησε. Ολοκληρώνοντας δε, θεωρούμε ότι το άνοιγμα της αγοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται σαν κίνδυνος για τους εργαζόμενους, αντίθετα για μια καλή ευκαιρία που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Για την ε, αναθεώρηση τώρα του κανονισμού για τα συμβόλαια με το δημόσιο 1370 του 2007, εκεί έχουμε αρκετές τροπολογίες αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε εμείς να τις υποστηρίξουμε σαν Επιτροπή. Θεωρούμε ότι για αυτά τα συμβόλαια από το δημόσιο βάση δημόσιων διαγωνισμών αυτός θα πρέπει να είναι γενικός κανόνας και η μελέτη επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση Επιτροπής το σημαντικό είναι να είμαστε αποτελεσματικότεροι με ε, θα στο 20-30% ε, όχι μόνο οικονομετρική ανάλυση επιτροπής αλλά αποτέλεσμα της πείρας που διαθέτουν τα κράτη-μέλη τα οποία προχωρούν σε αυτούς τους δημόσιους διαγωνισμούς ε, και ειδικότερα στη Γερμανία. Αυτό πέρα από αυτή την αποτελεσματικότητα των διαγωνισμών αυτών ε, θα πρέπει να τονίσουμε και τη διαφάνεια, τη σημασία της ε, στην ε, χρησιμοποίηση δημόσιου χρήματος, κάτι που θα πρέπει να διέπει, να χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή αγορά, τη δημόσια και γιατί εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εξαιρέσεις στον τομέα των σιδεροδρόμων. Ολοκληρώνω λοιπόν λέγοντας ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι όσες τροπολογίες θέλουν να αποδυναμώσουν, να καταργήσουν ένα σημεία ε, της πρότασης Επιτροπής και για τις δημοσίες, τη συμμετοχή δημοσίου δεν συμφωνούμε με αυτές. Βέβαια μια μεταβατική περίοδος επίσης για τις ε, αρμόδιους που να προσαρμοστούν στη νέα οργάνωση και για τις δημόσιες αυτές προσφορές αγορές, διαγωνισμούς. Ε, ε, λέμε ότι η προθεσμία θα μπορεί να είναι το 2019. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα άνοιγμα το 2029 γιατί θα επέτρεπε σε κράτη-μέλη να ε, αναθέσουν απευθείας έργα χωρίς διαφάνεια που θα οκληρώταν το 2044 τελικά και να, τελειώσουμε σχετικά με τα χαμηλή στιγμή συμβόλαια που μπορεί να ανατεθούν άμεσα, όπως λέει και η Επιτροπή, αυτό τα ελάχιστα 5 εκατομμυρίων ευρώ για 15 χρόνια, ας πούμε, μέχρι 70 τόσα εκατομμύρια ευρώ, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει αντιμεκίνηση βάση για να το πάμε από το 5 εκατομμύρια στο 10 εκατομμύρια ετησίως και για τη 2012-34 για την οδηγία αυτή η διαφοροποίηση των λειτουργιών σχετικά με την υποδομή και προμήθεια υπηρεσιών θεωρούμε ότι χρειάζονται ρυθμίσεις ώστε οι νέοι φορείς να μην ασκείται να μην διαφέρουν από τους ιστορικούς φορείς που δούλευαν πάντα εκεί. Χρειάζεται μια διαφάνεια και θεωρούμε ότι η πρότασή μας είναι πραγματικά εύκαμπτη, ευλίγιστη, γιατί τι προτείνει μια δομή κατάλληλη ανάμεσα σε αυτές τις δύο πτυχές με μια ολοκληρωμένη ταυτόχρονα σεβόμενη όμως κανόνες αυτό που λέμε συνοικοτήχος ε, Τώρα σχετικά με το άνοιγμα των εμπορικών υπηρεσιών που προβλέπεται στα πλαίσια της πρότασης αυτής, ε, όπως προβλέπει ο εισηγητής, ε, απαραίτητο είναι να διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα στις ε, δημόσια συμβόλαια και στα εμπορικά παρόμοια και τι προβλέπει ο εισηγητής στην πρόταση και στο νομοθετικό κείμενο να υπάρξει και μια σειρά λεπτομερών κριτηρίων ώστε να μπορέσουμε έτσι να δούμε αυτό το πλαίσιο το οικονομικό, το κείμενο το οικονομικό. Εάν δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα σχετικά με αυτά τα μέτρα, τότε δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται, ότι απαιτείται όλα αυτά να ενταχθούν στο κείμενο το νομοθετικό. Ήδη έχουμε μια εντολή στην πρώτη δέσμη των ε, συνδρομικών μέτρων για να προετοιμάσουμε αυτά τα πράγματα. Αυτό και κάνουμε άλλωστε. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να επιμείνω ιδιαίτερα. Τρέφω την ελπίδα ότι ο εισηγητής και τα μέλη της Επιτροπής θα προχωρήσουν για την οριστικοποίηση αυτής της έκθεσης και η Επιτροπή είναι στη διάθεση του εισηγητού και στα μέλη της Επιτροπής σας για να προσφέρουμε και συγκροματικές πληροφορίες. Ευχαριστούμε κύριε Λίζουα, ο Πρόεδρος. Και ολοκληρώνουμε τώρα. Ο εισηγητή άκουσες ε, πολλές ερωτήσεις. Ελπίζομαι να έχεις και πολλές απαντήσεις. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διαφορούς σκαιώδε και τις διάφορες ομάδες ε, για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Θα ήθελα επίσης να τους ευχαριστήσω για τα σχόλιά τους σήμερα το πρωί και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για την παρέμβασή της πρέπει να σας πω ότι δεν εκπλήσωμαι και ιδιαίτερα από τις διάφορες παρεμβάσεις που μένουν μέσα στις γραμμές που είχα αντιληφθεί όταν διάβασα και τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, εγώ Αισθάνομαι να υπάρχει σύγκληση με την ομάδα του ΕΛΚ και με την ομάδα των Πρασίνων και συγκεκριμένα τις τροπολογίες που κατατέθηκαν, καθώς ε, σε μεγάλο βαθμό και σύντομα θα τη σχολιάσω ανατροπολογία, αλλά σε μεγάλο βαθμό οι τροπολογίες ε, που καταθέσατε θα μπορούν να ενταχθούν σε συμβαστικές τροπολογίες και θα το συζητήσουμε αυτά τις επόμενες μέρες. Είναι σαφές ότι η προσέγγιση των φιλελευθέρων έρχεται σε αντίθεση με τη δική μας προσέγγιση, ακόμα και αν η είναι η της απασχόλησης και τη θέση των σιρουδοδρόμων ε, στα διάφορα μέσα μεταφορών. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου την πτυχή της ασφάλειας, που είναι ένα σημαντικό στοιχείο και θα πρέπει να έχουμε κατά νου και την πτυχή της προσβασιμότητας και ιδίω όταν ε, μιλάμε για περιοχές που ε, δεν ε, εξυπηρετούνται όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν ίσως να έχουμε κοινού στόχους μεν, αλλά δεν νομίζω ότι θα επιλέξουμε την ίδια οδό για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς δε. Έτσι λοιπόν, αυτά όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε και φυσικά είμαι ανοιχτός να ακούσω τα διάφορα επιχειρήματα και είμαι σίγουρος ότι κατά την εκπόνηση συμβιβαστικών τροπολογιών και των καταλόγων ψηφοφορίας θα είναι πολύ πλούσιες οι συζητήσεις μας. Ευχαριστώ, Φρεντερίκ. Λοιπόν, έχουμε το εξής ε, χρονοδιάγραμμα. Στις 14 ε, Νοεμβρίου θα συζητήσουμε τώρα για τις, τόσο για τις συμβαστικές προτάσεις ε, όσο και θα ψηφίσουμε στις 26 Νοεμβρίου ε, θα ψηφίσουν ε, στην Τραν ε, και κατόπιν θα ακολουθήσει μια ελπίζουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάμε στο επόμενο θέμα της μεσης το 14, που πρόκειται για το εξής. Πρόκειται για την κοινωνική διάσταση της ε, ΟΝΕ που δεν είναι εδώ παρούσα η συγγετρία γιατί μας εκπροσωπεί στο Βίλνιους αλλά δεν ξέρω μήπως ε, ε, θέλει κάποιος συνάδελφος να κάνει κάποια παρατήρηση έστω και αν δεν είναι εδώ παρούσα η κυρία Περές Παρακαλώ Ο Σάμπα Έρη έχει πρώτος το λόγο και μετά ο Φίλ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για το λόγο. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που μπορούμε να μιλήσουμε κάποιος πιο λεπτομερώς ε, για τα θέματα που τέθηκαν στην ψηφορία. Όταν ε, δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση της Κομισιόν, την καλωσορίσαμε και το πράξαμε καταρχήν, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη πως όταν ε, οικοδομούμε την ΟΝΕ και τους κανόνες θέλουμε να έχουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τον κοινωνικό αντίκτυπο αυτών. Επομένως, θέλαμε να έχουμε μια κοινωνική διάσταση στην ε, ΟΝΕ και υποστηρίζουμε βεβαίως την ιδέα αυτή και πιστεύουμε ότι είναι καλή ιδέα να έχουμε αυτό το scoreboard, ε, αυτό το πίνακα και αυτό αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Κομισιόν, όμως εδώ μιλάμε στο να δοθούν κάποιες δυνατότητες για να έχουμε μία πιο ακριβή εικόνα. Όμως είμαστε κατά του να εξαχθούν αυτόματα συμπεράσματα έτσι όπως αναφέρεται στο έγγραφο γιατί πιστεύουμε ότι το τομέα της κοινωνικής πολιτικής δεν επιτρέπει πολύ μεγάλη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε εθνικές στρατηγικές που ισχύουν και θα έπρεπε να δούμε και τους νομικούς περιορισμούς εδώ, να το αναλύσουμε αυτά για να δούμε ότι έχουμε τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές και αν δούμε τις κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης και το θέμα των δικτών συμμετοχής, ένταξης, τότε θα πρέπει να έχουμε μια ακριβέστερη ανάλυση γιατί αυτό αφορά και τα κράτη-μέλη, τους δίνει τροφή για σκέψη και καλές ιδέες. Όμως δεν θέλουμε αυτόματα συμπεράσματα να εξάγονται βάσει αυτής της κοινωνικής ανάλυσης όπως συνηθίζεται σε άλλους τομείς πολιτικής. Εδώ μιλάμε για κοινέ ευρωπαϊκές αρμοδιότητες από τη μία και εθνικές αρμοδιότητες από την άλλη. Επομένως, στο κείμενο έχουμε μία σειρά προβλημάτων και μία σειρά μετόπων. Θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες διαγραφές ή κάποιες τροποποιήσεις Νομίζω πάντως ότι θα υπάρχει μια ευκαιρία για μας να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ναι, το βρήκα. Καταρχήν θέλουμε να διαγράψουμε το σημείο F, το I, το X και θέλουμε να διαγράψουμε ένα τμήμα του σημείου 2 κτλ. τα Επομένως, Νομίζω ότι τώρα θα ήταν κρίμα να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες για να μην μακρηγορώ, δεν χρειάζεται, αλλά συνολικά θα έλεγα ότι πρέπει να απαντήσουμε εμείς στην ανακοίνωση της Κομίσιον και να πούμε ότι σεβόμαστε τις επιθυμίες των κρατών μελών ότι σεβόμαστε να μην αφαιρεθούν οι αρμοδιότητές τους όταν μιλάμε στην κοινωνική, για την κοινωνική πολιτική. Θέλουμε να σεβαστούμε τις βασικές συνθήκες και ξέρετε, αναφερθήκαμε στην οικοδόμηση μιας πολιτικής στρατηγικής. Θα πρέπει και το Κοινοβούλιο να διαδραματίσει το ρόλο του και θα πρέπει να ακουστεί η φωνή του. Θα θέλουμε να συνεργαστούμε με την Κομισιόν γι' αυτό. και αυτά θέλουμε να αντικατοπτρίζονται στο κείμενο. Αλλά προφανώς είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε με του και να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσαμπαόρη. Από το ΕΛΚ ο κύριο Σέρκα, από τους Yeah. Ναι. Πρόεδρε, ευχαριστώ είναι σημαντική αυτή τη στιγμή στην πολιτική συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα στο τέλος της θητείας μας και είναι νέο κεφάλαιο. Θα πρέπει να έχουμε αυτό το θάρρος, αυτό το όχημα να το οδηγήσουμε κοιτάζοντας ε, και μπροστά αλλά και από το καθρεφτάκι πίσω γιατί ουσιαστικά είναι μια νέα αρχιτεκτονική στην Ευρώπη για το μέλλον το συζητάμε και προτείνει η Επιτροπή δειλά-δειλά όμως η αρχιτεκτονική αυτή η καινούρια να μην λησμονήσει την κοινωνική διάσταση. Η νέα οικονομική νομισματική Ευρώπη έχει ήδη μια κοινωνική διάσταση. Δεν θα πρέπει να έχει μια κοινωνική διάσταση αλλά υπάρχει το έλλειμμα το χρέος, η μάχη για τη συνεργασία πάνω στις προκλήσεις τις μακροοικονομικές, αλλά το όλο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τίποτα, τι θα γίνει, τι γίνεται με τους πολίτες, τι γίνεται με την αγορά εργασία, τι συμβαίνει και ποιος είναι το μέλλον της στρατηγικής 2020 λόγω της κρίσης που εμφανίστηκε. Η ανακοίνωση της Επιτροπής λοιπόν ε, μετά από πολλές υποσχέσεις του Συμβουλίου και του Προέδρου Μπαρόσου που είπε ότι θα γίνει έχουμε όμως ε, μια εικόνα και πρέπει να πούμε εδώ να το καλωσορίσουμε αυτό γιατί είναι αυτό ε, η πρόταση της Επιτροπής που είναι επιθετική. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε το υλικό και στους υπόλοιπους συναδέλφους για την κοινωνική διάσταση. Σε επικοδομητικά λοιπόν να υπενθυμίσουμε στους συναδελφούς ότι ε, δεν συμμετέχει το Συμβούλιο τελικά. Εδώ θα πρέπει να συμμετάσχει όμως, γιατί όπως είναι λογικό θα πρέπει να έχει μια κοινοτική μέθοδο που να το χαρακτηρίζει και να είναι ανάμεσα στα τρία όργανα τη ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είπα και στον συναδελφό Όρη, γιατί είναι ιδιαίτερα αντιφατικό όταν μιλάμε ότι πρέπει να ακούσουμε αυτά που προβάλλονται από εθνικής ε, πλευράς δεν ακούμε το Συμβούλιο, τις απόψεις του Συμβουλίου για το μέλλον αυτής της αρχιτεκτονικής του πυλώνα του κοινωνικού. Θα το δούμε και προσεχώς και θα πρέπει και άντυπα να τους προσκαλέσουμε. Πέρα όμως από αυτό που συζητάμε τώρα για το ψήφισμα, τι γίνεται διαδικαστικά αυτό που συζητάμε τώρα όλοι, θα πρέπει να είναι ε, ε, κατοστοιχειώδες. Όχι για, συζήτηση, για την κίνηση, για τη συζήτηση αυτή και να λείπει το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη, έτσι. Αυτό λοιπόν, ελπίζω με τη σοφία σας εσείς να βρεθούμε μια λύση και υπάρχει όμως μια διαφορά, μια απόκληση μεταξύ μας. Ποιος θα πρέπει να είναι ο κοινωνικός πυλώνας. Να πω και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που η ουσιαστική ομάδα τα λέει αυτά, Εντάξει, καλωσορίζουμε αυτή την ανακοίνωση και επιτέλους κάτι έχουμε στα χέρια μας ώστε να ξεκινήσουμε την πορεία μας ε, αυτά τα κοινωνικά προβλήματα να τα θέσουμε στο ίδιο επίπεδο από οικονομικής πλευράς αυτό το εξάμεινο όπως ε, και τις προκλήσεις μαρκοοικονομικές και εμείς ε, θα προτείνουμε τροπολογίες για να ενισχύσουμε πράγματα που λέγονται ήδη εκεί μέσα. Σημαντικό πραγματικά είναι να πούμε ότι μας προσφέρει Επιτροπή ένα θέμα που είναι σημαντικό απαραίτητο, αλλά ε, συμπεριλαμβάνει δείκτες που θα πρέπει να δείξουν ε, την ε, έλλειψη ισορροπίας της κοινωνικής, γιατί ε, κάθε φορά, μέρα βέβαια που κοιτάζει κανείς τον καθρέφτη, να βλέπει τον εαυτό του πιο άσχημο και πιο γέρο. Και... Αλλά θα πρέπει όμως και να χρησιμεύει το καθεφτάκι για να διορθώνουμε τα προβλήματα. Εδώ έχουμε πέντε βασικά στοιχεία για να δούμε πώς έχει η κατάσταση. Αλλά λείπουν τα σημαντικά. Εμείς θα προτείνουμε σε αυτό το ψήφισμα μέρε τροπολογίες για να το ενισχύσουμε, για να μην λησμονηθούν η ε, φτώχεια ε, τα παιδιά, το ένα το άλλο και όλα αυτά, πώς έχουμε αυτές τις μαύρες τρύπες σε θέματα κοινωνικά στην Ευρώπη. Και το μεγάλο το πρόβλημα τώρα ποιο είναι, όχι μόνο να έχουμε μέσω σημαντικό ανάλυσης αλλά και τα στοιχεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν πολιτικές που να προλαβαίνουμε έτσι και μετά να διορθώνουμε. Το ίδιο ακριβώς όπως έγινε και με την έλλειψη ισορροπίας μακροοικονομικής. Θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε και να έχουμε τις δυνατότητες να προλαβαίνουμε τα προβλήματα και μετά να διορθώνουμε και όλος όταν εμφανίζονται και στην ανακοίνωση Επιτροπής. Αυτό λείπει γιατί είναι ιδιαίτερα απομακρυσμένοι από αυτό και με το Συμβούλιο του Επιτροπή ή με την έλλειψη ισορροπίας ε, κοινωνική ότι όλα αυτά παίζουν τεράστιο ρόλο στην κρίση στην οικονομική. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε με τις τροπολογίες μας. Θα τονίσουμε αυτό. Το προφανές ότι η οικονομική κρίση που οφείλεται βασικά στις διαφορές στην Ευρώπη και στο ευρώ παραλίγο να πεθάνει πέρυσι λόγω της έλλειψης συνεργασίας συμμετρίας γιατί με τη έλλειψη αυτής συμμετρίας δεν μπορούμε να έχουμε εσωτερική αγορά Ευρώπη αφού λειτουργούν τα πάντα διαφορετικά αποκλίνουν και κάθε μέρα στις βασικές παραμέτρους διαφέρουν πρέπει όμως να, να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη ναι, μια αγορά εργασίας ναι για τα εισοδήματα, ναι για τα φορολογικά αλλά όχι να συνεχίσουμε αυτές διαφόρες ε, και αντί να υιοθετήσουμε μια πολιτική συνοχής και σύγκλησης, ε, αντίθετα να απομακρυνόμαστε. Θα τονίσουμε λοιπόν τη σημασία αυτού γιατί διαφορετικά σε μερικά χρόνια θα ανακαλύψουμε ακόμα περισσότερα, πιο δραματικά. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα ενίο νόμισμα εάν η οικονομική πολιτική δεν είναι συντονισμένη και κατάλληλη. Θα τα δούμε σε μερικά χρόνια ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια παρόμοια πολιτική και αν δεν υπάρξει και μια κοινωνική πολιτική συντονισμένη με συνοχή και θα το δούμε έτσι. Βλέπουμε από εδώ και από εκεί διάφορα που προτείνονται για την ανεργία των νέων και να λένε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση προς το κέντρο από τις περιφερειακές χώρες. Πρέπει, έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι αυτό δεν γίνεται, δεν μπορούν να υποστηριχθούν έτσι με εργατικά χέρια που θα συγκλίνει προς το κέντρο και θα ε, καθίστανται ακόμα πιο φτωχές αυτές οι χώρες. Δεν μπορούμε να έχουμε φτωχή περιφέρεια και πλούσιο κέντρο. Έτσι, το μοναδικό μέσο, το φάρμακο, είναι να λάβουμε υπόψη μας τη σύγκληση, την κοινωνική, την περιφερειακή και όλες αυτές τις δυνατότητες. Αυτό είναι το βασικό. Όπως ο όροι που Κάπως τα είδε στενά τα πράγματα, με παροπίδες. Ε, όταν ακριβώς συζητάμε για τις τροπολογίες, θα πρέπει να το καταλάβει κανείς. Δεν είναι σοσιαλιστική η προπαγάνδα μας αυτά που προτείνουμε. Τίποτα δεν έχει καμία σχέση με τις εκλογές. Δεν ξέρουμε αν είναι και κανείς ε, υποψήφιος είναι το μέλλον της Ευρώπης, το μέλλον εκατομμυρίων και νέων και εργαζομένων. Να ξέρει κανείς τι θα γίνει, τα ίδια λάθη θα κάνουμε πάντα ή θα υποφεληθούμε από τη νέα αυτή διάσταση που μας προτείνει η ανακοίνωση Επιτροπής για πιο έξυπνη στρατηγική που θα μας επιτρέψει έτσι να σώσουμε την κοινωνική Ευρώπη. Από τη στιγμή που θα τη σώσουμε, την κοινωνική Ευρώπη θα σώσουμε και ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι. Λοιπόν, ε, τροπολογίες λογικές θα τις ε, συζητήσουμε με τους συναδέλφους. Όχι για δική μας προβολή της ομάδας μας, αλλά προσπάθεια όλων μας για να ξεφύγουμε από την κρίση και να είναι μια ευκαιρία για να βελτιώσουμε την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είναι πολύ λεπτά αυτά τα θέματα και πολύ σοβαρά και ίσως ε, θα μπορούσαμε όμως ε, να συντομεύσουμε γιατί έχουμε κάπως ε, καθυστερήσει, Φιλ. Δεν θα καθυστερήσω εγώ τόσο πολύ. Μικρόφωνο, παρακαλούμε. Συγγνώμη, έσβησε. Ναι, εδώ έχουμε ε, τον ε, σκιώδη να ευχαριστεί την ε, εισηγήτρια, αλλά όπως πιστεύετε, όπως τα αναμένετε, έχουμε κάποια θέματα με την πρόταση. Όπως και σε προηγούμενη συζήτηση δεν συμφωνούμε με τους αυτόμετους σταθεροποιητές, ούτε υποστηρίζουμε το μηχανισμό πυροδότησης. Επίσης, έχουμε προβλήματα με το ORT με αυτά τα εκτιμώντας και τα καθέσουμε τροπολογίες τουλάχιστον για τις παραγράφους 1, 2, 6, 10 και 16 και συμφωνούμε ότι μπορεί να υπάρχει καλύτερη παρακολουθήση των κοινωνικών δικτών και πιστεύουμε ότι οι κοινωνικοί δείκτες έχουν ένα ζωτικό ρόλο στο να συμπληρώσουν τους οικονομικούς δείκτες ε, αλλά Τώρα εδώ μπερδεύουμε τους οικονομικούς ε, και τους κοινωνικούς δείκτες σε ένα πίνακα της και νομίζω ότι ε, όλα αυτά είναι ανοησίες ε, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να παρουσιάσει οποιοδήποτε τελικό αποτέλεσμα θέλει. Και τι θα κάνει με αυτό το τελικό αποτέλεσμα τελικά κανείς. Εγώ νομίζω ότι η ιδέα του να έχουμε ένα τέτοιο μεικτό πίνακα αποτελεσμάτων δεν στέκει. Θα πρέπει να έχουμε κοινωνικούς δείκτες που να μπορούμε να τους εμπιστευτούμε και να τους κατανοήσουμε. Και αν μπορούμε να το πράξουμε αυτό, τότε θα μπορέσουμε να σημειώσουμε και πρόοδο. Έτσι λοιπόν, ο Φίλιππ ανυπομονεί για τη συζήτηση αυτή και τη συνεργασία επί του φακέλου αυτού τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλοι και εφόσον μίλησαν οι φιλελεύθεροι, τώρα θα δώσω το λόγο στους ε, ε, πράσινους. Ίσως θα μπορέσω να φέρω λίγο ε, ευκρίνεια σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Αυτά που είναι σαφή είναι ότι το ευρώ χρειάζεται μια οικονομική διακυβέρνηση. Η ιδέα δεν είναι να πούμε ότι τα κοινωνικά θέματα πρέπει να συζητώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που ενδιαφέρει είναι όπως συμβαίνει και στην νομισματική πολιτική, όπου όλα γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι ότι ό,τι αποφασίζεται ε, ισχύει για όλη την Ευρώπη. Να υπάρχει όμως μια ισορροπία ε, και εδώ στηρίζω τον Αλεσάνδρο έτσι ώστε να μην ε, διολιστήσουμε σε μία λάθος κατάσταση ε, και αυτό αφορά μια πλούσια χώρα γιατί αυτή η λάθος κατάσταση αφορά όλους. Περί αυτού πρόκειται. Εμείς λοιπόν οι πράσινοι θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν αυτόματα συστήματα εξισορρόπησης. Αυτό δεν υπάρχει στην έκθεση Κομισιόν. Πρόκειται για μακροοικονομικά εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι είναι πολυσχηδής, να είναι μια σταθερή ένωση. Και τα εργαλεία που υπάρχουν δεν αρκούν. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι πρόβλημα. Το ότι όλο και περισσότερο δημιουργείται ένα άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Γι' αυτό πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε πέρα από τα εθνικά σύνορα να μεριμνήσουμε η ανεργία και η φτώχεια να μην λαμβάνουν υπερβολικές διαστάσεις σε μια χώρα γιατί αυτό βλάπτει όλες τις χώρες και τις πλούσιες σε τελική ανάλυση όλοι υποφελούνται από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά την άποψή μου αυτή είναι η προσπάθεια της ε, Κομισιόν ε, και γι' αυτό χρειαζόμαστε το ψήφισμα. Πρέπει λοιπόν να μεριμνήσουμε έτσι ώστε όλοι αυτοί οι τομείς της οικονομικής ε, διακυβέρνησης να ρυθμίζονται σε επίπεδο αρμοδιοτήτων. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν βέβαια οι μέθοδοι για να κατίστανται δυνατά ορισμένα πράγματα. Η μέθοδος είναι ο συντονισμός, όπου τα κράτη-μέλη λαμβάνουν μια απόφαση για το scoreboard, για τα κριτήρια. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά εκείνοι που προτείνουν αυτά τα θέματα και που μεριμνούν έτσι ώστε να υπάρχουν στην σε διάταξη του Συμβουλίου, αυτοί είμαστε εμείς. Ακριβώς αυτό κάναμε και με την εγγύηση των νέων. Και αυτό δεν είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι απόφαση των κρατών μελών ε, κυρίως για θέματα συντονισμού. Αυτή είναι η ουσία του θέματος και νομίζω ότι αν συνεργαστούμε επ' αυτού του θέματος τότε θα προχωρήσουμε πολύ και νομίζω ότι αυτό θα εξυπηρετήσει κυρίως εκείνα τα κράτη τα οποία υποφέρουν τώρα περισσότερο από την κρίση. Γιατί και αυτά δεν μπορούν να βγουν μόνο τους από το βούρκο, χρειάζονται την αλληλεγγύη μας. Την αλληλεγγύη τη χρειάζεται ολόκληρη η Ευρώπη και αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να βγούμε από την κρίση. Σε ευχαριστούμε πολύ Ελίζαμπετ. Ε, για λόγους ε, χρόνου δεν θα μιλήσω εγώ. Ο κύριος ε, Σάμπα έχει το λόγο για δύο μόνο λεπτά. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, να πω μερικά πράγματα στον Αλεχάνδρο. Είναι κάπως αργά να έχουμε μια συζήτηση τώρα με το Συμβούλιο. Ίσως να βρούμε μια λύση. Θα είχαμε όμως να έχουμε μια διαφορετική βάση για τη συζήτηση αυτή. μην θέτουμε, μην υποβάλουμε ερωτήματα ενώ γνωρίζουμε τις απαντήσεις. Εάν υποβάλουμε ερωτήσεις, τότε θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε και άλλους στόχους. Όχι, δεν λέω αυτά για τους σοσιαλιστές. Θα πρέπει να επωφεληθεί κανείς από όλες τις ε, δυνατότητες που προσφέρονται. Εντάξει, σήμερα, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της φτώχειας, του αγώνα κατά της φτώχειας. Γι' αυτό θα πρέπει να δείξουμε μια σοβαρή στάση συζητώντας για το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πάρα πολλά μέσα, πάρα πολλά εργαλεία, περισμένα βέβαια, αλλά όσον αφορά την περιφέρεια έχουμε τα διορθωτικά ταμεία, μην το ξεχνάμε, και όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ναι μεν δεν διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά χρήματα και ότι τα χρήματα αυτά δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα όλα για να βοηθήσουν και το συντονισμό της αναλύσεις, τη συλλογή εμπειριών και όλα αυτά να δημοσιευθούν. Δεν μπορούμε να λύσουμε έτσι εύκολα τα προβλήματα αυτά στη θέση των κρατών μελών και δεν μπορούμε να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πετύχει λύσεις σε θέματα κοινωνικών πολιτικών. Θα πρέπει να υποβάλουμε προτάσεις. Εμείς είμαστε εταίροι. Εταίροι για την εξέβρεση λύσεων. Αλλά θα πρέπει να αποφεύγουμε πορείες και προσανατολισμούς που δεν εξυπηρετούν σε τίποτα και που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα ταμεία δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνηση αυτόματους μηχανισμούς γιατί δεν έχουμε τα μέσα. Πρέπει όμως ε, τα κράτη να προσέξουν ποια είναι τα προβλήματα και αυτό γίνεται από τη στιγμή που ξεκινάμε πρωτοβουλίες υπέρ των νέων. 6 ε, εκατομμύρια αφιερώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό, αλλά είναι μια σταγόνα στον ωκεανό και θα πρέπει να, λάβουμε, να λάβουμε, αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να ενθαρρύνουμε. Αλλά τα κράτη-μέλη πρέπει να πληρώσουν τα έξοδα. Αυτή ήταν μια συζήτηση που σίγουρα θα τη συνεχίσουμε. Οι τροπολογίε μέχρι τις 23 ε, Οκτωβρίου, 12 η ώρα, παρακαλώ μόνο στα αγγλικά, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για γραπτή μετάφραση και στις 5 ε, Νοεμβρίου ε, θα εξετάσουμε τόσο τις ε, τροπολογίες και θα ψηφίσουμε, όσο και θα ψηφίσουμε. Αυτά για το 14. Πάμε στο 15 τώρα παρακαλώ. Πρόκειται για την κοινωνική προστασία για όλους και για τους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους. Η κυρία Μπλινκεβιτσούτε έχει το λόγο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το ότι μπορεί κανείς να συντάξει μία έκθεση στην Επιτροπή μας για την κοινωνική προστασία για όλους και τους ε, ε, εργαζόμενους που εργάζονται Εδώ είναι πολύ σημαντικό, σημαντικό να μιλάμε για το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως σε αυτά τα πλαίσια από τη στιγμή που υπάρχουν περικοπές στον προπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα η ανεργία αυξάνεται ο ηλεγγυοδός και σε κοινωνικές παροχές και βλέπουμε τον προϋπολογισμό από την άλλη μεριά που αντιμετωπίζει τρομερές περικοπές. Μείωση των εισοδημάτων, αύξηση της ανεργίας, λοιπόν μείωση των ε, κρατήσεων και αυτό απειλεί και δυσκολεύει το κοινωνικό πρότυπο το ευρωπαϊκό. Βέβαια εδώ με την έκθεση αυτή καλύπτονται πολλές πτυχές. Το πρώτη κύρια για την κοινωνική ασφάλιση για όλους και η δεύτερη πτυχή έχει να κάνει με τους αυτόνομους εργαζόμενους και την ασφάλισή τους. Θα σας πω σύντομα ποιες, ποια είναι τα κύρια σημεία τα οποία εμφανίζονται στην έκθεση αυτή. Είναι απαραίτητο, τονίζω, να αναπτύξουμε και να εξυγχρονίσουμε το σύστημα κοινωνικής προστασίας και αυτό για να την εξασφαλίσουμε κατάλληλα για όλους, με πρόσβαση για όλους και να μην γίνεται καμία διάκριση βάρος κανενός και να μπορεί κανείς όμως και να αντιδράσει κατάλληλα στην δημογραφική ε, αύξηση αυτή και να επέμβουμε στην αγορά εργασίας. Ε, Χρειάζεται χρηματοδότηση και υπεύθυνη και αηφόρος στα πλαίσια μιας κρίσης. Ε, και αυτό για τις κοινωνικ... μέσω κοινωνικών κατάλληλων παροχών. με τις επενδύσεις αυτές τις κοινωνικές μπορούμε να πετύχουμε στόχους κοινωνικούς. Γι' αυτό αυτές οι κοινωνικές επενδύσεις, θα πούμε έτσι, δεν είναι δαπάνες, είναι επενδύσεις πραγματικά. Προσκαλώ λοιπόν τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν την εξέβρεση θέσεων εργασίας για τους νέους, να καταβάλουν προσπάθεια και να μην υπάρξει καμία διάκριση εις βάρος των νέων εργαζομένων και να μην ε, είναι και τα δικαιώματά τους περιορισμένα. Θα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία και στους πιο ευαίσθητους, ευάλωτους, τους άνεργους, ε, του ανάπηρους, νέες οικογένειες, όλους αυτούς θα πρέπει να προστατευτούν κοινωνικά αυτές οι κατηγορίες με τις κοινωνικές κατάλληλες παροχές. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσέξουν ώστε να υπάρξει καλύτερη πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές, κυρίως σε εκείνους που είναι περισσότερο ευάλωτοι και για εκείνους που χρειάζονται φροντίδες ε, μακροπρόθεσμα. Προσέξτε λοιπόν το θέμα της πρόσβασης σε κοινωνικές, πρασ... Ε, σε κοινωνικές παροχές στις αγροτικές περιοχές γιατί υπάρχουν, ε, υπάρχει μια εκμετάλλευση εργαζομένων πολύ συχνά. Γι' αυτό να δώσουμε τη μάχη μας κατά της παράνομης εργασίας ε, που δεν τη δηλώνουν οι εργοδότες για καλύτερη κοινωνική προστασία αυτών των εργαζομένων. Και επίσης να τονίσω κάτι, ε, όταν γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης δεν γίνονται οι συνήθεις βασ αντί για αυτές να έχουμε μη συνήθεις νόμιμες ε, σχέσεις εργασίας και θα πρέπει να δούμε τον κανονισμό για τον συντονισμό ε, για την προστασία την κοινωνική. Και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάω να κάνει μια ανάλυση της καταστάσεως και να σιγουρευτεί ότι οι τροπολογίες, οι τροποποιήσεις μάλλον στο εργατικό δίκαιο από εθνικής πλευράς να μην επηρεάσουν αρνητικά την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων και η κοινωνική αυτή ασφάλιση, το δικαίωμα σε αυτή να μην παραβιάζεται. Και κάτι ακόμα για τους αυτόνομους εργαζόμενους, γιατί, γιατί αποδίδω στην κατηγορία αυτή ιδιαίτερη σημασία στην έκθεση. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε μερικούς κινδύνους, αρκετούς κινδύνους. Η φύση απασχόλησης αλλάζει, όλο και περισσότερο αυτόνομοι εργαζόμενοι υπάρχουν και ο κίνδυνος είναι οι ομάδες αυτές εργανομένων να μην προστατεύονται κοινωνικά κατάλληλα. Και γίνεται πιο δύσκολη πολιτική απέναντι σε αυτούς τους εργαζόμενους επειδή δεν υπάρχει σαφή συγκεκριμένος ορισμός αυτών των αυτόνομα απασχολούμενων ε, Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ ζητάω από την Επιτροπή να επεξεργαστεί ένα ορισμό σαφή, συγκεκριμένο, ώστε να μπορεί κανείς να ξέρει ακριβώς ποιες είναι αυτές οι μορφές εργασίας, οι αυτόνομοι εργαζόμενοι κλπ. Γιατί με τον τρόπο αυτό και μόνο θα μπορέσουμε σωστά να εφαρμόσουμε αυτές τις κοινωνικές εγγυήσεις και να γίνουν σεβαστά τα κοινωνικά δικαιώματα. Θα πρέπει να δούμε κατάλληλα επίσης και τους ψευδοαυτόνομους ε, γιατί αυτό θα είναι, είναι, είναι το μέσο για θέμητο ανταγωνισμό και ταυτόχρονα και δικαιολογία ώστε ορισμένοι εργαζόμενοι να μην ε, μπορούν να κάνουν χρήση των νόμιμων δικαιωμάτων τους. Άρα λοιπόν εμφανίζεται κίνδυνος για ντάμπιν κοινωνικό στρέβλωση του ανταγωνισμού και παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων. Να τονίσω για μια ακόμα φορά τις σημαντικότερες πτυχές από την δεν υπάρχει κοινό ορισμός. Καθιστά αυτό πιο δύσκολο ακόμα τον συντονισμό σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση των αυτόνομα απασχολουμένων και ε, ουσιαστικά μια περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και δεν υπάρχουν και αρκετά στοιχεία για αυτούς τους αυτόνομα απασχολούμενους και γι' αυτό χρειάζονται να ενημερώσουμε τα στατιστικά στοιχεία, να είναι και περισσότερο λεπτόμερη για να μπορέσουμε έτσι να προσέχουμε και μάλιστα αποτελεσματικότερα τις οικονομικές δραστηριότητες των διαφόρων ομάδων αυτών των απασχολουμένων και να κάνουμε την κατάλληλη ανάλυση ανάλογα με το φύλλο του, την ηλικία του, την κοινωνική του θέση κλπ. Και επίσης θα πρέπει να προσέξουμε ώστε οι περιπτώσεις εκείνες που έχουν να κάνουν με προχωρημένη ηλικία, είτε με αναπηρία, είτε με ε, την άδεια ε, πατρότητας, όλα αυτά να μην παραβιάζονται και χρειάζεται όλα αυτά να ενημερώνονται υποχρεωτικά, όλοι αυτοί θα πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνονται για αυτά τα δικαιώματά τους λόγω της θέσης τους, όπως και για άλλα δικαιώματά τους, αλλά και υποχρεώσεις τους λόγω της θέσης τους. Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εγγυώνται παρόμοια ενημέρωση. Παρακαλώ προσέξτε και μια ακόμα κατηγορία, όλο και περισσότερο πολυάριθμη εργαζομένων, αυτόνομα απασχολούμενων που είναι οικονομικά εξαρτώμενοι. Λόγω της φύσης εργασίας τους είναι σχεδόν μισθωτοί. Γι' αυτό λοιπόν τα κοινωνικά τους δικαιώματα θα πρέπει να είναι συγκρίσιμα με εκείνα των μισθωτών. Δεν έχω όμως χρόνο σχεδόν άλλο στη διάθεσή μου, σε αυτά θα αρκεστώ και περιμένω τις ε, παρατηρήσεις ε, των συναδέλφων ε, και του συγητού και ελπίζω με τις παρεμβάσεις αυτές να βελτιώσουμε την έκθεση. Πολύ ωραία. Ε, έχουμε τους εξηγητές ε, των Φιλιππέγγεων μετά η Μαρή, η κυρία Κορνέλισεν και μετά κάποιος από την Επιτροπή. Φιλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι η μετάφραση στα αγγλικά δεν ήταν διαθέσιμη μέχρι χθες το απόγευμα και είχαμε τριμερή διάλογο χθε ε, το απόγευμα. Έτσι λοιπόν ε, πραγματικά είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν ένας-δύο τομεί που μπορώ να σχολιάσω. Τα επίπεδα της ε, πρόσβασης στην κοινωνική ασφάλιση Ακόμη και αν ε, κατάλληλα τα θέματα αυτά, πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά, είναι καλό να έχουμε μία συζήτηση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επίσης, συμφωνώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν πρακτικά βήματα για την καταπολέμηση της, ε, του κοινωνικού αποκλεισμού και χαίρομαι που αναγνωρίζει η συγκεντρία τις διαφορές ε, στις πρακτικές των κρατών μελών. Επίσης, ε, συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι η αυτοποσχόληση μπορεί να είναι μια θετική μορφή ευελιξίας της αγοράς εργασίας, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλα επίπεδα κοινωνικής προστασίας. Αναρωτιέμαι αν η Κομισιόν θα μπορεί να μας δώσει κάποιο νομικό ορισμό, μπορούμε να τη ρωτήσουμε, να τη το ζητήσουμε, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί πολλά από αυτά σχετίζονται με τους φορολογικούς νόμους ε, και κώδικες σε διάφορες χώρες, γιατί επειδή αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών μπορεί να υπάρχει πρόβλημα και να μην έχουμε ένα κοινό ορισμό που να καλύπτει την φορολογική κατάσταση σε κάθε χώρα. Και επίσης ε, δεν νομίζω ότι είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν ε, να ε, επιβάλλει κυρώσει στους εργοδότε. Θα πρότεινε η Κομισιόν να προτείνει κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ για τα κράτη-μέλη σε αυτό το τομέα. Αυτά έχω εξετάσει μέχρι τώρα. Αλλά ανυπομονώ να συνεργαστώ επικοδομητικά με την εισηγήτρια τη επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ κύριε Κορνέλισεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση αυτή τη στιγμή γιατί σε καιρούς κρίσης ε, όχι μόνο είδαμε αύξηση των αυτοπασχολούμενων, αλλά άλλαξε και το κινητρό τους να εργάζονται σε αυτοπασχόληση. Πάντοτε πιστεύαμε ότι οι άνθρωποι διάλεγαν την αυτοπασχόληση λόγω της ελευθερίας που τους έδινε και την δυνατότητα για καινοτόμη εργασία. Όμως, ε, πολύ περισσότεροι έχουν γίνει τώρα αυτά γιατί αναγκάζονται, γιατί οι εργοδότες δεν είναι πρόθυμοι να προσλάβουν με μια κανονική σύμβαση. Και επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια μείωση στις δομές φροντίδας για τα παιδιά και αυτό έχει ανάγκασε τις γυναίκες να γίνουν αυτοπασχολούμενες, να καθορίζουν ε, το χρόνο και τον τόπο εργασία τους. Και έχουμε φυσικά και πολλούς κινητούς εργαζομένους. Παίζουμε τους χάρη ε, ε, ε, η αυτοπασχόληση επιτρέπει την εκμετάλλευση των εργαζομένων και στις χώρες που εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια μέτρα μεταβατικά έναντι των ανατολικών χωρών ε, το χάρη δική μου χωρί, λενδιά έχει αποφασίσει να λάβει κάποια μέτρα έναντι των Κροατών που θα έλθουν ως εργαζόμενοι αυτοαποσχολούμενοι και αυτό τους κάνει ευάλωτους στην εκμετάλλευση. Έτσι λοιπόν, έχοντας κατά νου όλα αυτά, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τρόπους για να τα διορθώσουμε όλα αυτά και ε, κυρίως να σκεφτούμε ότι οι αυτοαπασχολούμενοι είναι η νέα κατηγορία φτωχών σε πολλά κράτη-μέλη. Εγώ συμφωνώ κύριε Μπένιον ότι μπορεί να έχουμε κάποια εμπόδια και θα πρέπει να ορίσουμε τους αυτοπασχολούμενους και να ορίσουμε και τον εργαζόμενο. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση λαμβάνει χρόνια εδώ και δεκαετίες. Επίσης, στα πλαίσια της κινητικότητας, ε, ίσως ε, θα ε, μπορούσαμε να δούμε τον ορισμό της αυτοπασχόλησης έτσι όπως ορίζεται στο κράτος υποδοχής, για να καταστήσουμε λιγότερο δυνατή την εκμετάλλευση. Ούτε εγώ μπόρεσα να δω το κείμενο λεπτομερώς, αλλά φυσικά υπομονούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση με την εισηγήτρια και τους κοιόδης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρή. Από την Κομισιόν υπάρχει κάποιος. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, γιατί ούτε εμεί είχαμε καιρό να μπούμε στι λεπτομέρειε τη έκθεση. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά σημεία επί των οποίων συμφωνούμε ότι η κοινωνική επένδυση είναι επένδυση, αλλά ε, έγινε και ένα σχόλιο για τι δυσκολίε εξέβρεση ενό κοινού ορισμού. Εδώ θα ήθελα να πω ότι φυσικά βλέπουμε ότι έχουμε παράνομη εργασία και μια ψευδής κατάσταση ε, αυτοαπασχολούμενο αποτελεί μια συνέπεια της προβληματικής νομοθεσίας. Όμως θα συνεχίσουμε όλη αυτή την εργασία και συνάδελφοι θα επανέλθουν με περισσότερες λεπτομερίες για τη δράση που ήδη αναλαμβάνουμε. Όμως θα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά σε διάφορους κανονισμούς και πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, εισηγήτρια, για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπενιόν. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι είναι τα κράτη-μέλη αυτά που είναι υπεύθυνα για την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία, όμως και εμείς είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα κυρίως ε, στα πλαίσια μιας κρίσης και ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης τα ευάλωτα άτομα είναι αυτά που έχουν πληγεί περισσότερο και γι' αυτό πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να ποινικοποιεί τους πιο ευπαθείς, τους πιο ευάλωτους. Ο κύριος Μπένιον, η κυρία Κορνέλισεν και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφεραν ε, το θέμα των ορισμών. Είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε ένα κοινό ορισμό για να γίνεται κατανοητός σε όλα τα κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε ίσως να σκεφτεί βάσει ποιων κριτηρίων θα μπορούσαμε να έχουμε έναν κοινό ορισμό. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που κυρία Κορνέλισεν παρουσίασε την αποψή τη στην Επιτροπή ΦΑΜ και αναφέρθηκε ιδίω στην κοινωνική προστασία των γυναικών. Αυτό είναι κάτι πολύ επίκαιρο σήμερα και νομίζω ότι όλοι εμείς συνεργαζόμενοι από κοινού στην Επιτροπή Απασχόλησης θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μία έκθεση πολύ σημαντική για το Συμβούλιο και για την Κομισιόν, για όλους. Εγώ είμαι έτοιμη να εργαστώ από τους συναδέλφους. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο κατατίθενται οι τροπολογίες μέχρι τις 24 Οκτωβρίου και μέχρι τις 24 Νοεμβρίου θα εξετάσουμε το θέμα και το Δεκέμβρη θα εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να γίνει αυτή η συζήτηση στην Επιτροπή ε, Απασχόλησης κανονικά μετά το 15, έχετε το 16, προηγουμένως όμως είχαμε αλλάξει την ημερήσια διάταξη. Τώρα έχουμε το 13 που είναι πώς μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δημιουργία φιλόξενου περιβάλλοντος ε, για τις μικρές και μεγάλες επιχείρησεις κτλ. Αντρέα Μακιντάρα, έχετε το λόγο. Χαίρομαι που συμφωνα η Επιτροπή μας για να παράξουμε αυτή την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Ήδη είχαμε δύο γνωμοδοτήσεις για το τομέα αυτό. Η μία αφορούσε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η άλλη αφορούσε τη μείωση της γραφειοκρατίας. Και έχουμε λάβει πλήρη υποστήριξη από αυτή την Επιτροπή και για τα δύο αυτά θέματα. Νομίζω ότι όλοι κατανοούμε πω η επασχόληση είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και ελπίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Όπως ε, ξέρετε, οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις και πολύ μικρές ε, επιχειρήσεις παρέχουν 90 εκατομμύρια θέσεων εργασίας και αυτό είναι τεράστιο δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για την ανάπτυξη και την καινοτομία και καθώς το 85% των ε, νέων ε, θέσεων εργασίας ε, τα τελευταία 10 χρόνια ήρθαν από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις. Προσπάθησα να αντιμετωπίσω στην έκθεση αυτή έχω διαιρέσει σε διάφορους τομείς όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, ε, η επιχειρηματικότητα και οι δεξιότητες. Και στο θέμα αυτό νομίζω ότι μας ενσυχεί ιδιαίτερα ότι ο αριθμός των πολιτών που θέλουν να είναι αυτοπεσχολούμενοι μειώθηκε από το 45% στο 37% τα τελευταία τρία χρόνια. Φυσικά και η προηγούμενη συζήτηση αναφέρονταν στο θέμα αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό το επιχειρηματικό πνεύμα ε, να προωθείται από πολύ μικρή ηλικία και ήδη από το πανεπιστήμιο και να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουμε κάποιον να ξεκινήσει μια επιχείρηση και να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε ορισμένε περιπτώσεις όπου έχουμε κάποιους έντιμους επιχειρηματίες που ίσως ε, δεν τα, πέτυχαν στην πρώτη δεν τα κατάφεραν στην πρώτη τους απόπειρα. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον επίσης αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, για το REFIT που έρχεται από την Κομισιόν, το πρόγραμμα αυτό. Και οι κύριες προτάσεις, η ε, πραγματική εστίαση για το REFIT θα πρέπει να είναι στην απλούστευση προτάσεων όπου θα είχαμε πραγματική επίπτωση στη μείωση του αχθούς για τις επιχειρήσεις. Νομίζω πρέπει να καλωσορίσουμε όσο έχει κάνει η Κομισιόν μέχρι τώρα. 5.500 νομικές απαιτήσεις έχουν καταργηθεί τα τελευταία χρόνια και έχουμε εξοικονομήσει 27 εκατομμύρια λίρες περισσότερα σε ευρώ και την επόμενη εβδομάδα ανυπομονούμε να ακούσουμε τις προτάσεις του κυρίου Μπρέσο για την περικοπή των κανονισμών της υπερβολικής νομοθεσίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο ο Πρωθυπουργό ε, θέσπισε μία task force για τι επιχειρήσεις που θα εκπονήσει μία έκθεση με στόχο να πιστεί την προσοχή σε κάποιους επαχθεί κανόνες ε, που ουσιαστικά παρεμποδίζουν ε, την ανταγωνιστικότητα των βρετανικών επιχειρήσεων και θα αναφερθεί και σε κάποια θέματα για τους εξαγωγείς, τις startups και όσους αναπτύσσουν νέα προϊόντα. Ο Πρωθυπουργό επίσης απέφθηνε έκκληση και σε άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για να λάβουν μέτρα να μειώσουν την περίτη νομοθεσία όταν θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα και νομίζω ότι είναι πολύ ευπρόσδεκτη αυτή η πρωτοβουλία. Έχουν εκφράσει άποψη κάποιοι επιχειρηματίε, οι οποίοι λένε ότι καλέ είναι οι ιδέες αλλά μπορεί να χαθούν στο δρόμο της εφαρμογή και αυτό μπορεί να έχει πολλές επιζημίες συνέπειε. Πόσο συχνά το έχουμε ακούσει αυτό. Επίσης, το συνέστημα ότι την εντύπωση ότι οι μικρές επιχειρήσεις θίγονται δυσανάλογα, πλήττονται δυσανάλογα από την γραφειοκρατία. Εγώ ήμουν πολύ ικανοποιημένη που είχαμε μία ακρόαση στην Επιτροπή αυτή πριν να εκπονήσω αυτή την έκθεση. Στην ακρόαση εκείνη ακούστηκαν διάφορες ε, οπτικές και απόψεις και νομίζω ότι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα που μερικές φορές είναι και κάπως επίμαχο είναι το θέμα της ασφάλειας και της υγείας και θέλω να το ξεκαθαρίσω όπως έγινε και στην ακρόαση. Εδώ θα έπρεπε να στοχεύουμε στο να μειώσουμε τη γραφεία, όχι το επίπεδο της προστασίας των εργαζομένων και πράγματι αν μειώσουμε την πολυπλοκότητα και μπορούν πιο εύκολα να σεβαστούν τους κανόνες οι μικρές εταιρείες, ε, τότε ε, προστατεύουμε καλύτερα και τους εργαζομένους μας. Ε, φυσικά υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών απόψεων για το πώς θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα θέματα της ανεργίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και ελπίζω να μπορούμε να συνεργαστούμε σε ένα καλό πνεύμα συνεργασίας και να βρούμε τη χρυσή τομή. Και Φυσικά θα υθετήσω στο δυνατό περισσότερα σχόλια. Είναι δυνατόν, ανυπομονώ, να συνεργαστώ με τους κοιόδης για την εκθεσία αυτή και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταθέσουμε κάποιες συγκεκριμένε προτάσεις που τα κράτη, μέλη, κομισιών και επιχειρήσεις θα μπορούσαν να υθετήσουν. Ευχαριστώ. <clears throat> Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τους ε, σκιώδης έχω την Μαρή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Μακεντάιρ. Ε, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις για να ξεκινήσουν και είναι πολύ σημαντικό για εκείνες να αποκτήσουν τις ε, σωστές ε, πληροφορίες έτσι ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση ε, στην πίστη, στη χρηματοδότηση. Βεβαίως έγινε αναφορά στην ευελικτή αγορά εργασίας, αυτό δεν με εξέπληξε καθόλου και παρότι υπάρχουν αρκετά θέματα με τα οποία συμφωνούμε όπως παραδείγματος χάρη να μάθει κανείς περισσότερα στη δουλειά και να περιορίσει την ε, γραφειοκρατία πρέπει να υπάρχει κάποιο σύστημα εξορροπήσεων και ελέγχου γιατί και κάποια θέματα γραφειοκρατικά δεν είναι παντελώς άχρηστα νομίζω ότι το να μάθουν οι νέοι πάνω στην θέση εργασίας αυτό τους βοηθάει για να αποκτήσουν εμπειρία και ε, με τον τρόπο αυτό δεν γίνονται και τόσο θύματα της ε, εκμετάλλευσης ε, για αυτήν η εργασία. Σας είπα λοιπόν ότι θα προτιμούσα να υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου και ελέγχων και εξισορροπήσεων και ελπίζουμε τελικά να καταλήξουμε με μια καλή έκθεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γκουτιέρες είναι ο σκιώδης εκ μέρους των σοσιαλιστών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο Σέρτζο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτή η έκθεση έχει πολλές ελλείψεις, ε, δεν γνωρίζει τα πράγματα για μας τις μικρομεσαίες, ε, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Λοιπόν, αυτό που έλεγε και η κυρία Κορνέλης, ναι, όπως επίσης και το κοινωνικό κόστος και τις ε, αγορές εργασίες. Θα πρέπει να δούμε πώς θα το υποστηρίξουμε. Θα έχουμε δυσκολίες αν δεν διορθώσουμε τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αυτές οι δαπάνες σημαίνουν μεγάλο μέρος του κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά μέχρι πέντε φορές αναβάζεται το κοινωνικό κόστος ε, των μισθών αλλά τι γίνεται με το ενεργειακό κόστος ε, που αντιμετωπίζουν πολλές ε, εταιρείε όπως και το κόστος μισθών αμοιβών και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη έχουν ένα σταθερό κόστος ε, και βέβαια τους μισθούς αλλά ε, μια σωστή αμοιβή για τους εργαζόμενους είτε για την ανεργία είτε για τις συνταξιοδότηση. Υπάρχει ένα πρόβλημα αυτό για να δημιουργήσουν ε, θέσεις απασχόλησης παρά το κόστος το άλλο που λέμε. Και εδώ αυτό είναι κάπως λανθασμένη σαν γραμμή. Και ε, πώς ε, συμφωνήσω με την συγγήτρια ότι θα πρέπει να δούμε και πάλι τα πρότυπά μας για να μην έχουμε γραφειοκρατία. Τι σημαίνει όμως αυτό, αναφέρεται στην όλη συζήτηση και όπως λέγεται στην Επιτροπή, τι γίνεται, δεν είναι μόνο διαφορά ερμηνείας, αλλά και προθέσεων και περιεχομένου. Όταν ακριβώς θέλει κανείς να βγάλει από τη μέση την γραφοκρατία και πώς να βελτιώσει τα πράγματα, να στουστεύσει ε, των ΜΕΤ, των όσων χρειάζονται για την σύσταση, για, την, ε, ε, για μια καινούργια εταιρεία ανάλογα με το μέγεθής της θα πρέπει να έχουμε κάτι το συγκεκριμένο όμως τη στιγμή που θα θέσουμε επιτάπητος προτάσεις γιατί αν μιλάμε έτσι γενικά στην οδηγία για το χρόνο εργασίας για την ασφάλεια, για την προσυνεργασία και να ζητάμε ευκαμψία ή απορρίθμιση Αυτά που ζητάμε εμείς οι ζωλιστές δεν είναι αυτά που ακριβώς ε, ε, θα πετύχουμε. Αντίθετα ανοίγουμε πόρτες για απορρίθμιση έτσι και είναι μια απαγορευτική γραμμή την οποία εμείς δεν θα ανεχθούμε. Και ορισμένα κενά τα οποία δεν εμφανίζονται σε αυτό το σχέδιο και που θα μπορούσαμε να τα επεξεργαστούμε, να ασχοληθούμε μαζί εδώ σε όλη την Ευρώπη μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρώτο που σου ζητάνε και πρώτο που λένε ότι έχουν ένα πρόβλημα χρηματοδότηση, δεν έχουν πιστώσεις κυρίως στις νότιες χώρες, είτε ότι η πίστοση, τα δάνεια είναι ακριβά σε σχέση με άλλους ε, από άλλες χώρες. Αυτό το πράγμα δεν εξετάζεται γιατί αυτές οι λίγες πιστώσεις, οι, οι φτηνές πιστώσεις ε, δίδονται στις μεγάλες ε, εταιρείες, μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στις μικρομεσαίες. Έχουμε πρόβλημα ακριβώς ε, χρηματοδότησης, δεν αντιμετωπίζεται και δεν γίνεται καμία αναφορά σε αυτή την ε, πρωτοβουλία πριν από μερικούς μήνες ας πούμε ένα μέρος ε, της εγγύησης για τους νέους να χρησιμοποιηθεί εν μέρει ακριβώς για μια πίστοση για καλύτερες ε, συνθήκες για την εργασία των νέων κυρίως σε χώρες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα ανεργίας είτε ένα κατάλληλο business program για δημιουργία επιχειρήσεων. Θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα των μικρομεσαίων για κοινοτομίε. Είναι εκτό προγραμμάτων για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά του. Αυτό είναι απαραίτητο για το μέλλον να το βελτιώσουν αυτό και να δούμε και το κόστο βέβαια των αμοιβών και αφήνουμε απ' έξω πολλές μορφές νέας οικονομίας που είναι, θα απασχολήσουν στο μέλλον την ε, ευρωπαϊκή οικονομία και την κοινωνική οικονομία για τα υπόλοιπα εντάξει αλλά αυτό μας απασχολεί μας απασχολεί τον ε, πρόβλημα το δίθεν αυτόνομα απασχολουμένων επειδή δεν υπάρχει δουλειά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες υπάρχει μια όθηση εκείνη που από μακρύ χρονικό διάστημα αναζητούν εργασία και προσπαθούν να το βρουν αυτό μέσω μιας κατάλληλης ε, αυτόνομης απασχόλησης. Τι γίνεται και υπάρχουν και άλλοι που αποκλείονται από τις επιχειρήσεις ε, και αναφέρονται σαν αυτόνομοι. Δεν θέλουν να είναι αυτόνομοι όμως ε, αλλά ουσιαστικά έχουν αποκλειστεί από την αγορά εργασίας και προσπαθούν έτσι να γλιτώσουν κόστος οι εταιρείε αυτές. Υπάρχει αυτό το ε, πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή εδώ είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το πρόβλημα και να προσπαθήσουμε να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις. Ολοκληρώνω λοιπόν ε, βλέπω να υπάρχουν κενά ορισμένα στην όλη έκθεση και ορισμένα θέματα που είτε αντιμετωπίζονται διαφορετικά και διαφορετικά η ομάδα μας ε, δεν θα μπορούσε να τα υποστηρίξει. Χρειάζονται προσπάθειες για να επιληθούν. Ευχαριστούμε πολύ Στέτζο και έχω άλλους δύο που έχουν ζητήσει το λόγο. Ο Φιλ Μπένιεν εκ μέρους των Φιλελευθέρων και ο Σάμπα Έρη για το ΕΛΚ και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και μετά η εισηγήτρια θα κλείσει αυτή τη συζήτηση. Οφείλει έχει το λόγο. Κοιτάξτε και εδώ ε, πρόκειται πάλι για τον κύριο Ντεμπάκερ που είναι σκιοδησηγητής. Ε, Δυστυχώ πήρε την έκθεση λίγο πριν φύγει για το Ταλίν. Ε, έτσι λοιπόν ε, τα σχόλια του είναι κυρίω αυτά που θα ήθελε να περιλαμβάνει η έκθεση. Συμφωνεί λοιπόν ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι η ραχοκοκαλιά τη οικονομία μα, ότι πρέπει να βελτιωθούν οι δυνατότητε για ένα επιχειρηματία για να μπορεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Θέλει επίση να επισημάνει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην προκύψει απλά άλλη μια έκθεση για τις ε, μικρομεσαίες, ενώ κατ' ουσίαν δεν αλλάζει τίποτα στην πρακτική. Επίσης ε, ήταν ε, ο εισηγητής σχετικά με την βελτιωμένη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, κάτι που παρουσιάστηκε στις αρχές του έτους και η Κομισιόν παρουσίασε μια έκθεση για την επιχειρηματικότητα. Μέχρι τώρα βλέπουμε οι επιχειρηματίες να διαμαρτύρονται ότι δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Άρα δηλαδή έχει έρθει πια στιγμή για δράση και όχι πια για λόγια. Νομίζω ότι στην έκθεση πρέπει να προσέξουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες και αναφέρει τέσσερις τομείς ε, προτεραιότητων. Καταρχήν, βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, όχι βραχυπρόθεσμα μέτρα, αλλά πραγματικά μεταρρυθμίσεις. Ε. Δεύτερον, στο σύστημα εκπαίδευσης αναφέρει ότι χρειαζόμαστε ε, εκπαιδευτικό σύστημα υψηλού επίπεδου, όπου οι καθηγητές έχουν ειδικά προσόντα, τα συστήματα έχουν προσαρμοστεί στα απαραίτητα προσόντα. Παράλληλα, πρέπει να εντάσσεται και η επιχειρηματική πραγματικότητα στο υπάρχον σύστημα. Να μειωθεί το διοικητικό άχθος ε, για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην αρχή και αργότερα. Επίσης, ε, η νομοθεσία δεν θα πρέπει να επιβάλλει ε, ιδιαίτερη επιβάρνηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να υπάρχει λοιπόν ευελιξία στην αγορά εργασίας και ένα δίκτυο ασφαλείας, να ενθαρρύνονται περισσότεροι να μπουν στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι απαραίτητο για να έχουμε ε, εργατικό δυναμικό με προσόντα. Αν δεν υπάρχει αυτό, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν και να αναπτυχθούν. Ο Φίλιπ προσβλέπει στο να συζητηθεί αυτό το θέμα κατά τις επόμενες επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο τελευταίος ομιλητής εκ μέρου των Ευρωβουλευτών, ο κ. Σαμπαέρη. Ευχαριστώ. Δεν θα μακρηγορήσω, απλώς ε, θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Μπουλάν είναι ο δικός μας ε, εισηγητής ε, και δεν λέμε ότι δεν θέλουμε να πάρουμε το λόγο, αλλά υπάρχουν ψηφοφορίες και σε άλλες επιτροπές αυτή τη στιγμή και πρέπει να πάμε εκεί είπε ο κ. Μπουλάν ότι θα προσπαθούσε να επιστρέψει, δεν τα κατάφερε. Αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα, το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ε, και φυσικά θα συνεισφέρουμε στην όλη συζήτηση. Πολύ ωραία. Εκ μέρου τη Επιτροπή η κυρία Ολίβους. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν καλωσορίζει την έκθεση αυτή, αυτή η οποία επικεντρώνεται σε πολύ σκόπιμα ζητήματα, πώ μπορεί να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τις startup για τη δημιουργία θέσεων είναι στο επίκεντρο τη ε, της βιομηχανικής πολιτικής μας. Εδώ τονίζονται θέματα όπως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η πρόσβαση στην αγορά και δεξιότητες που είναι κάποιοι από τους πυλώνες της στρατηγικής μας. Οι μικρές και μισές επιχειρήσεις είναι ζωτικές για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υιοθέτησε η Κομισιόν το σχέδιο δράσης για την επιχειρηματικότητα προκειμένου να έρθουν τα εφιστάμενα εμπόδια και να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη για την καλύτερη νομοθεσία. Ακολουθεί η Κομισιόν μια ενεργητική συνέχεια για τον την κατάργηση των 10 ε, πλέον επαχθών νομοθετημάτων για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Επίσης, ε, είχαμε τον Οκτώβριο μία ανακοίνωση όπου η Κομισιόν αναφέρει ανατομία πολιτικής που θα αναλάβει περαιτέρω δράσεις για την απλούστευση, την απόσυρση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι είναι πιο εύκολη η εφαρμογή της νομοθεσίας. Ο κύριος της Κομισιόν είναι να υπάρχουν αυτές να διευκολύνουμε τις εξελίξεις στην αγορά, επιταχύνοντας την υιοθέτηση νέας τεχνολογίας και τα εμπόδια για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Ό,τι αφορά τον ενεργό ρόλο των επιχειρήσεων και τη δέσμευσή τους είναι πάρα πολύ σημαντικά για να υπάρχει δημιουργία θέσεων και πάλι στην Ευρώπη. Επικεντρωνόμαστε στην ικανότητά μα ε, να έχουμε τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς για να τα πετύχουμε τις δράσεις αυτές και σε εθνικό επίπεδο και συμπεριλαμβάνουν και διαφορετικών μεταρρυθμίσεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και τονίζεται και από αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση η συγκήτρια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης. Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σου. Ξέρω ότι υπάρχουν τομεί όπου έχουμε διαφωνίες, αλλά είναι υπομονώ να λάβω τις προτάσεις σου και τις τροπολογίες σου. Κατόπιν, για τα όσα είπε ο κύριος Γκουτιέρες Πρέτο, ναι, έχει κάποιες ελλείψεις η έκθεση και θα ήθελα να δω κάποιες τροπολογίες. Ε, ήταν πολύ χρήσιμο αυτό που είπατε για το θέμα της ενέργειας, όμως πρέπει να σκεφτείτε ότι εδώ μιλάμε και για ένα περιορισμό, μόνο έξι σελίδες ε, ε, μπορεί να περιλαμβάνει μια έκθεση δίας πρωτοβουλία. Εγώ θα τροποποιήσω την έκθεσή μου, σας διαβεβαιώ. Όμως υπάρχει η παράγραφος 13 που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Αν ε, θέλετε να συμπληρώσετε, ευχαρίστως. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το Φιλ και τον κύριο Ντεμπάκερ για το ενδιαφέρον τους. Περιμένω και τις δικές σας τροπολογίες και τον κύριο Όρη, εκ μέρους του κύριου Μπουλάν. Ευχαριστώ την ε, υποστήριξή σας και το ενδιαφέρον σας. Νομίζω ότι η δική μας Επιτροπή μπορεί να κάνει τη διαφορά θέτοντας ε, από κοινού όλες αυτές τις πτυχές σε μια έκθεση και έτσι μπορούμε να προσθέσουμε και τη δική μας φωνή στη φωνή άλλων που ασκούν πίεση στην Κομισιόν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία πτώνησα ήταν οι διαφορές ε, στο πόσες μέρες χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια επιχείρηση και την πολυπλοκότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαι πολύ καρμμένη που μιλάμε μόνο για 13 μέρες, ενώ στη Μάλτα 40. Έτσι λοιπόν θα ήταν καλό αν μπορούσαμε να έχουμε την ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών, έτσι ώστε όλοι να βελτιωθούν. Και θα κλείσω λέγοντας ότι η δημιουργία των επιχειρήσεων για τη μείωση της ανεργίας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Χθες στη δική μου περιφέρεια έγινε μια ανακοίνωση ότι δημιουργήθηκαν 13.000 θέσεις εργασίας το τελευταίο τρίμηνο και μειώνεται ε, το ποσοστό της ενεργείας. Εγώ αυτή την προσέγγιση θα ήθελα να δω παντού στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει μια διορία 4 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε λοιπόν πρέπει να έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες και κατόπιν ε, θα ψηφίσουμε εδώ το Δεκέμβρη και ενδεχομένως αν χρειαστεί και τον Ιανουάριο. Ο κύριος Χάουιτ ε, τώρα μπορεί να λάβει το λόγο, αλλά παρακαλώ να είστε σύντομος, Ρίτσαρτ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και για την ευελιξία που δίνετε. Όπως ξέρετε, το θέμα αυτό που συζητάμε είναι ένα θέμα ε, το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ από κοινού με την εταιρική ευθύνη. Αυτά είναι προϋποθέσεις ε, για τη διαφάνεια σε μια εταιρεία ε, Πάντως ε, θέλω να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις στο Κοινοβούλιο ε, με όλες τις πολιτικές ομάδες και έχουμε στηρίξει την αρχή ότι πρέπει να αλλάξουν ε, οι οδηγίες για εταιρικό δίκαιο έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Αυτή ήταν μια σύσταση αυτής της Επιτροπής πέρυσι και ο κ. Μπανιέ προς τιμήν του δημοσίευσε μια σχετική πρόταση και εσείς ε, ως ε, Επιτροπή με ορίσατε ως εισηγητή και σας ευχαριστώ πολύ. Έχω καταθέσει μία σειρά ε, τροπολογιών. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Οι πρώτες αφορούν στην αλυσίδα προσφοράς και την αλυσίδα που έχει σχέση με την αξία. Τα μέλη της Επιτροπής θα κατανοήσουν ότι αν μια έκθεση περιορίζεται απλά στις λειτουργίες των κεντρικών γραφείων ε, στο φιλοξενούμενο, στο κράτος που φιλοξενεί την εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό δεν είναι σωστό γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές ευθύνε που αφορούν ολόκληρη την αλυσίδα. Μπορούμε βέβαια να περάσουμε και στην άλλη, στο άλλο άκρο να πούμε ότι μια εταιρεία πρέπει να ξέρει τους πάντες μέσα σε αυτή την αλυσίδα τροφοδοσίας. Το θέμα είναι ότι έχει διαπιστωθεί στην πράξη πρακτική, στην πράξη ότι οι εταιρείε ε, γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται και ε, επιδεικνύουν την δέουσα επιμέλεια. Τώρα, κατά πόσον θα ονοματίσουμε τα διεθνή πλαίσια, ε, εδώ δίστανται οι απόψεις. Εγώ στηρίζω την άποψη ότι πρέπει να γνωρίζουμε το πλαίσιο, πρέπει να είναι γνωστό το πλαίσιο. Βέβαια να μην γίνουμε πολύ αυστηροί στις τροπολογίες μου λέω ότι πρέπει να αλλάξουν ονομασία οι διάφορες οδηγίες που υπάρχουν και επίσης ε, και οι οδηγίες που αφορούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτά τα έχω βάλει με τη σειρά που σας τα ανέφερα και έχω για κάποια υποσημείωση. Και με τον τρόπο αυτό ε, δίνουμε ένα μήνυμα χωρίς να είμαστε νομικά δεσμευτικοί. Ελπίζω να με στηρίξετε σε αυτή μου την τροπολογία. Επίσης στηρίζω, προτείνω, με συγχωρείτε, να στηρίξουμε μια υποχρέωση εφαρμογής. Αλλά να πούμε στα κράτη-μέλη, βέβαια, το πώς θα γίνει αυτό εναπόκειται σε εσά. Και ελπίζω επ' αυτού να συμφωνήσει η Επιτροπή. Αν θέλετε αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, συστήνω και προτείνω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ε, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές στα χρηματοψηφιακά. Υπάρχουν τέτοιες οδηγίες, δεν είναι βέβαια δεσμευτικές. Επειδή εδώ πρόκειται για την έκθεση περί ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβάλλοντος, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε αυτό που σας πρότεινα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ορισμένα από τα θέματα που προτείνουν οι επενδυτές, οι εκθέσεις ε, ε, ψηφίζονται σε γενικές συνελεύσεις των εταιριών και αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Προέρχεται βέβαια από τους επενδυτές και πρέπει να τη λάβουμε την πρόταση ε, σοβαρά υπόψη μας. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, πολύ ευχαριστώ να απαντήσω ε, σε ερωτήσεις. Ξέρετε όλοι σας ότι εγώ στηρίζω την έννοια της ολοκληρωμένης έκθεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν μπορεί σήμερα να αποφασίσει από αυτού. Είναι μια κίνηση που θα προχωρήσει στο μέλλον. Ε, το όλο θέμα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε δεν είναι τόσο η κοινωνική πολιτική, η επιπτώση στο περιβάλλον και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίσως εδώ να μην υπάρχουν οικονομικές προεκτάσεις, υπάρχουν όμως τελικά κάποιες και επιτιμούμε αυτό να το κατανοήσουν οι επιχειρήσεις και να το συμπεριλάβουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Υπάρχουν κάποιες εταιρείε που είναι πρωταθλητές σε αυτό. Θέλω βέβαια να το προχωρήσουμε όλο αυτό να υπάρχει ένα εδάφιο που να παραπέμπει στην οδηγία και να λέει ότι καλούμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία με έναν τρόπο ε, που θα είναι συνεπής ε, με αυτό που αποκαλούμε integrative reporting, ολοκληρωμένες ε, εκθέσεις. Αυτά είχα να πω και προσβλέπω στο να ακούσω και τις ε, απόψεις άλλων και ενδεχομένως και ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ε, Δύο έχουν στήσει το λόγο, ο Φίλιπ και ο Τόμας Μαν. Φίλιπ, είσαι ο πρώτος. Ε, Ευχαριστώ. Πάλι είναι από τον κύριο Ντεμπάκερ. Διάλεξε καλή μέρα να πάει στο Τάλιν, γιατί περισσότερες εκθέσεις του σήμερα συζητούνται. Πιστεύει ότι οι ευκαιρίες για την κοινωνική ευθύνη μπορούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Έτσι λοιπόν να είναι καλό να είναι ορατό το CSR στις εταιρείες. Ρωτά γιατί μόνο λιγότερο από το 10 της από τα 10% των αποκαλύπτουν πληροφορίες σε τακτική βάση. Αυτό γιατί δεν είναι πεπισμένε για την πρόσθετη θέμενη αξία θα πρέπει όμως να είναι σε αυτό ότι θα πρέπει να γίνεται σε κούσια βάση υποβολή εκθέσεων CSR για το διοικητικό άχθος. Ε, είναι πολύ κανομένο με το ότι ξερούνται οι μικρές και μεσέ επιχειρήσει Δεν είναι ότι δεν ωφελούνται από το CSR, αλλά ίσως να μην έχουν επαρκεί ε, ανθρώπινους πόρους και μπορεί να τους κοστίζει περισσότερο. Επίση, ο Φίλιπ καλωσορίζει την πρόταση τη Κομισιόν για το ότι δίνει ευελιξία στις εταιρείε, αλλά μπορεί να ε, σκεφτούμε ότι πρέπει να το εξηγήσουμε καλύτερα. Επίσης για την ευελιξία θέλει να τονίσει ότι πρέπει να αποφύγουμε το gold plating για κάποια κράτη-μέλη και χρειαζόμαστε ίσως κανόνες για όλα τα κράτη-μέλη και ανεπομονή να συζητήσει αυτό το φάκελο με, τους, ε, με τον συγητή στο μέλλον. Σε ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα ε, να πω κι εγώ κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ο Ρίτσο το ξέρει αυτό, δουλεύουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το θέμα της εταιρική ευθύνη και στο τέλος καταλήγαμε πάντα σε συμβαστική πρόταση και ελπίζω ότι θα το κάνουμε και πάλι αυτό. Όσον αφορά το θέμα της ε, του προαιρετικού ημί. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι ε, καταστήσαμε την εταιρική ευθύνη ως ένα σημαντικό στοιχείο του επιχειρηματικού πολιτισμού, της επιχείρησης απλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλές επιχειρήσεις ασχολούνται με την εταιρική ευθύνη και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως είναι και ένα δείγμα ανταγωνιστικότητας. Μπορεί μια εταιρεία να το προβάλλει αυτό. Ε, Δηλαδή, αν ας πούμε μια εταιρεία φέρει ευθύνη, αναλαμβάνει ευθύνη για την κοινωνία, για τους εργαζόμενους, για το πώς χειρίζεται το θέμα των πρώτων υλών, ε, αν τα χειρίζεται όλα αυτά καλά, είναι καλό και να το προβάλλει. Ε, Ρίτσαρτ, στην τελευταία σου έκθεση δεν ε, τοποθετήθηκες στο αν αυτό θα είναι υποχρεωτικό ή όχι οι εταιρείες θα πρέπει καταρχήν να προσαρμοστούν, όχι βέβαια οι μεγάλες, γιατί αυτές έχουν εμπειρογνώμονες και μπορούν να το κάνουν πολύ πιο εύκολα, αλλά οι μικρομεσαίες και δεν χρειάζεται για αυτές να δημιουργήσουμε γραφειοκρατικά εμπόδια. Απλά και μόνο το γεγονός ότι για την εταιρική ευθύνη έχουμε κάνει τόσα πολλά και λέμε σε εταιρείε να γίνεται πιο συγκεκριμένες, ήδη με αυτό ε, πετύχαμε πάρα πολλά. Είμαι σύντομος γιατί ξέρω ότι έχουμε καθυστερήσει. Ε, δεν ξέρω αν κάποιος από την Επιτροπή επιθυμεί να λάβει το λόγο. Από ό,τι βλέπω κανείς. Όχι, δεν θέλει κανείς. Πολύ ωραία. Ο Ρίτσαρτ ε, έχει το λόγο. Εσύ ξεκίνησε και εσύ θα τελειώσεις. Καταρχήν συμφωνώ ότι θα πρέπει να βρούμε ένα συμβασμό. Έχεις δίκιο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και επίσης για να είμαι σαφής, οι τροπολογίες που έχω καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής συνάδουν απόλυτα με όσο συμφωνήσαμε πέρσι. Είναι λοιπόν οι ίδιοι συμβασμοί για τα ίδια θέματα και έτσι θα ξεκονομήσουμε πάρα πολύ χρόνο και ευχαρίστως να συναντηθώ κατηδίαν με τους συναδέλφους για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά τη διατύπωση που χρησιμοποιούμε, όπως και πέρσι, εγώ κάνω έκκληση τώρα να μιλάμε ε, για δηλαδή ότι ε, δεν χρειάζεται να συμμορφούνται οι επιχειρήσεις, να μην το λέμε voluntary εκούσιο, όμως ξέρετε στα Ηνωμένα Έθνη είχε γίνει μια ολόκληρη συζήτηση που υιοθετήθηκε και από την Κομισιόν και λέει ότι πρέπει να υπάρχει ε, ουσιαστικά ένα μείγμα, να μην μιλάμε για voluntary έναντι του mandatory, του εκούσιου του υποχρεωτικού. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι και δικές σας επιφυλάξεις ε, και όχι μόνο οι δικέ σας, ξέρω ότι εκπροσωπείτε και μια ανησυχία που υπάρχει, είναι καλύτερα μέσω της διαδικασίας της συμμόρφωσης να διατυπωθεί. Και αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι χθε είχαμε μια σύσκεψη διαβούλευση υπό την ηγεσία της κυβέρνησης της Δανία και ε, μιλούσαμε για την ε, υποβολή εκθέσεων σε σχέση με την νομοθεσία αυτής της συμμόρφωσης και το 90% των εταιριών επιλέγουν να συμμορφωθούν, δεν τους αναγκάζει κανείς, αλλά το επιλέγουν γιατί έτσι φάνηκε ότι αυτό το είδος υποβολή εκθέσεων μπορεί να είναι καλό και για το περιβάλλον και για την κοινωνία αλλά και για τις επιχειρήσεις. Και έτσι λοιπόν ε, θέλω να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους προς αυτή την κατεύθυνση και είπες ε, και εσύ Τόμας ότι η Norvardisk ε, αυτή η μεγάλη ε, εταιρεία ήρθε σε αυτή την επιτροπή και υποστήριξε την προσέγγιση μας. Έτσι λοιπόν πολλοί από την επιχειρηματική κοινότητα μας υποστηρίζουν και είπε και κάποια πράγματα ο Φιλ, καταρχήν για το πεδίο εφαρμογή και τον αποκλεισμό των μικρών και μέσων επιχειρήσεων. Συμφωνώ απόλυτα γι' αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αλυσίδα εφοδιασμού για να υπάρχει μια θετική επιρροή στις μικρότερες επιχειρήσεις, όμως δεν νομίζω ότι μεγάλες εταιρείες πρέπει να κυρώνουν συμβόλαια ή να προσπαθούν ε, να μετακινούν τους δικούς τους κινήτους. Νομίζω ότι πρέπει να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βρούμε και το σωστό τρόπο πώς θα κινηθούμε έτσι ώστε να μην ε, πλήττονται οι μικρές επιχειρήσεις ε, και για το gold plating συμφωνώ απόλυτα. Θα δώσω ενθάρρυνση και στον αδελφό, αλλά και σε όλους μας ότι εδώ μιλάμε ότι αυτή η υποβολή εκθέσεων θα γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει συζητηθεί αυτό το θέμα και σε παγκόσμιο επίπεδο και το σχετικό έγγραφο έχει οθετηθεί από 6.000 εταιρείε παγκοσμίω. Έτσι λοιπόν εδώ δεν προωθούμε ένα δικό μας μόνο ευρωπαϊκό πρότυπο. Υπάρχουν οι δείκτες επίδοσης επί των οποίων πρέπει να αναφέρουν, να υποβαλούν εκθέσεις οι εταιρείε και υπάρχουν και διεθνή πρότυπα. Απλώς εδώ θέλουμε να τα προωθήσουμε βοηθήσουμε. Και αυτό είναι ο τρόπο πρόθεσή του και νομίζω ότι είναι η σωστή προσέγγιση και γι' αυτό την υποστηρίζω. Ευχαριστώ. Vielen Dank, ähm, Richard. Wir haben die Deadline für unsere Anträge bis zum 4. Μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, 12 η ώρα, είναι η διορία για τις ε, τροπολογίες. Ε, θα μιλήσουμε στις 5 Νοεμβρίου και στις 25 και θα ψηφίσουμε στις 26 Νοεμβρίου. Μετά έχουμε την Επιτροπή Γιούρη που είναι η κύρια Επιτροπή και μετά το Φεβρουάριο θα έχουμε την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Πάει λοιπόν το 19 και πάω τώρα πίσω στο σημείο 16. Ελίζαμπετ Μωρόν ε, Σατιέ θα ήταν εδώ, αλλά δεν είναι. Ο κύριος Σαμπαρούρη θα την αντικαταστήσει. Ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, ζητάει συγγνώμη η Ελίζαμπετ γιατί είναι στην εκλογική της περιφέρεια που υπάρχει εκεί μια συνάντηση και απαιτείται να είναι παρούσα. Δεν είναι ιδιαίτερα μπερδεμένη η έκθεση αυτή. Είναι ένας κανονισμός του Συμβουλίου 1800 μάλλον συγγνώμη του 2006 1800. 83. Ο Ιόλ ε, συνέταξε μία. Ο κ. ε, θα ήθελε να εκφράσει την άποψη του γι' αυτό και υποστηρίζεται η γνώμη του Κοινοβουλίου εδώ για μια συμπληρωματική στήριξη που αποφασίστηκε από τον Ιούλιο την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής από τους ε, ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων. Πρόκειται για ζημιές λόγω της κρίσης και μία αντιστάθμιση 84 εκατομμύρια τη Γαλλία, για την Ιταλία 25 εκατομμύρια και για την Ισπανία 17 εκατομμύρια κονδύλια που θα δοθούν στις χώρες αυτές. Και για την ανεργία των χώρων αυτών είναι υψηλότερη από ό,τι ο μέσος όρος ο κοινοτικός. Και οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων θεώρησαν ότι πρέπει να βοηθηθούν αυτές οι χώρες λόγω των ζημιών που υπέστησαν. Άρα λοιπόν με την έκθεση Ολμπριχτ ε, από τη στιγμή που συμφωνεί κανείς δεν ε, υπάρχει διάθεση για μεταβολές, δεν θα πρέπει να καθυστερήσουμε, θα πρέπει τα μέτρα αυτά να εφαρμοστούν, να ισχύσουν όσο γίνεται συντομότερα και η Ελίζαμπετ ε, υποστηρίζει την έκθεση της Περιφερειακής Επιτροπής χωρίς τροπολογίες, χωρίς προσθήκες. Τώρα, αν κάποιος θα ήθελε κάτι να προτείνει, μπορεί να το κάνει μέχρι τις 22 και 7 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σίγουρο αυτό το χρονοδιάγραμμα. Επόμενος ο μιλητής, ο Αλεσάνδρο, δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι άλλο. Πρόεδρε, όχι, απλώς θέλω να πω ότι η ομάδα των σοσιαλιστών δεν θα καταθέσει καμία τροπολογία. Συμφωνεί με την Ελιζαμπέτ ε, και αυτά πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου για να τεθούν σε εφαρμογή τα προγράμματα και οι σοσιαλιστές συμφωνούν με την συγκήτρια, δεν θα παρουσιάσουμε καμία τροπολογία. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Οι άλλοι όμως που θέλουν να καταθέσουν τροπολογίες πρέπει να προσθέσουν, γιατί όπως είπε και ο Σάμπαχ, η διορία είναι 22 Οκτωβρίου, 12 η ώρα, αλλά μόνο στα αγγλικά, γιατί ε, δεν έχουμε χρόνο, ίσως και να μην θέλετε και τροπολογίες. Στις 5 Νοεμβρίου θα εξετάσουμε το θέμα. Σάμπαχ, ε, και άλλη μια φορά θα λάβεις το λόγο και για το 17 που κανονικά θα ήταν στην άλλη κόζα, αλλά θα το παρουσιάσει εσύ Πρόκειται για την στρατηγική σχετικά ε, με την υλοποίηση των προγραμμάτων της περίοδου 7-13. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Να είναι στο εξωτερικό όλη τη βδομάδα ο κύριος Κώσα. Δεν μπορεί να παρευρεθεί εδώ, αλλά μου ζήτησε να διαβιβάσω τα κυρία μηνύματα που θα ήθελε να πει σε σχέση με το θέμα αυτό. Η πολιτική συνοχής Τη Ευρωπαϊκής Ένωση ε, για την περίοδο που αναφέρεται είναι αυτό που μας απασχολεί. Υπάρχουν δύο εκθέσεις, η έκθεση 7 και η έκθεση 8 της Κομισιόν και αυτές εξετάζουμε Τώρα, οι δύο εκθέσεις καλωσορίζονται από τον Άντα και θεωρεί ότι πρέπει η έκθεση για το 2014 να εξετάσει το μικροπρόθεσμο αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης ε, για οποιαδήποτε μείωση της συνοχής μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μείωση συνοχής, αυτό το κενό, αυτό το χάσμα που φαίνεται να ανοίγεται. Υπάρχουν ε, διάφορα προβλήματα όπως άνθρωποι που εγκαταλείπουν ε, το σχολείο και υψηλό ποσοστό τέτοιων μαθητών σε κάποιες περιφέρειες. Ε, επίσης πρέπει να δούμε αυτό το στόχο του 10% και πρέπει να δούμε πώς οι νέοι θα έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να μπουν στην αγορά εργασίας και ξέρουμε ότι η έλλειψη προσόντων συχνά οδηγεί σε ενεργεία και κατόπιν σε φτώχεια. Πρόσφατα ακούσαμε τον Επίτροπο να αναφέρεται στα συμπεράσματα που πρέπει να εξαχθούν από μία ανάλυση και ε, είχαν, είχαμε ήδη κάποιες αρνητικές προοπτικές ε, σε ό,τι αφορά την έβρεση της συνεργασίας από ανθρώπους που έχουν χαμηλή εξειδικευσή και πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Επίσης τονίζεται ότι σε ορισμένες περιφέρειες ε, η ανεργία παραμένει κάτω από το 16% εδώ και δεκαετίες είδαμε να υπάρχουν προβλήματα στο εσωτερικό κάποιων κρατών μελών, δηλαδή σε ορισμένες περιφέρειες έχουμε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης. Αυτό που πρέπει να κάνουμε στην Ευρώπη είναι να δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Αν μπορούμε να πληρώνουμε τις δημόσιες υπηρεσίες μας και αν θέλουμε να μπορούμε να τις χρηματοδοτούμε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις κοινωνικές πολιτικές, με το σύστημα συνταξιοδότησης, το σύστημα υγείας. Πρέπει να τα καλύπτουμε όλα αυτά. Και αν το δούμε και το θέμα από περιφερειακή σκοπιά, υπάρχουν σοβαρά μειονεκτήματα και υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο στο οποίο φυσικά την προσοχή μας, ένα λεγόμενο παράδοξο αστικό όπως το αποκαλεί. Αν δούμε τους δείκτες μπορεί να σχηματιστεί εντύπωση ότι κάποιες αστικές περιοχές μπορεί να φαίνεται ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι είναι στην πραγματικότητα. Έτσι και εδώ λοιπόν ε, βλέπουμε ανέχεια και σε αυτές τις μεγάλες πόλεις παρόλο που βρίσκονται σε οικονομικά αναπτυγμένα κράτη. Εξακολουθούν να υπάρχουν οικογένειες ε, με χαμηλή εντατικότητα εργασίας, μονογονικές οικογένειες, άνθρωποι που είναι κοντά στην ηλικία συνταξιδότησης, άνθρωποι που ζουν μόνοι τους και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε όλες αυτές τις ομάδες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι έχουν ισότιμες ευκαιρίες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και να άρουμε τα εμπόδια πρόσβασης ε, στην εργασία. Επίσης, ο Άνταμ έχει ερευνήσει το πώς μπορούμε να έχουμε συγκρίσιμους δείκτες, έτσι ώστε να μπορούμε να λάβουμε υπόψη τις δημογραφικές προκλήσεις ο Άνταμ ε, θα ήθελε να συνεργαστεί δημιουργικά με τους συναδέλφους ε, και να συμπεριλάβει επικοδομητικές τροπολογίες στο κείμενό του. Θα επανέλθει την επόμενη εβδομάδα, έτσι λοιπόν ε, θα ήθελε να τα συζητήσει όλα αυτά με τους συναδέλφους και σας ευχαριστώ εκ μέρους του. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλο ευρωβουλευτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να λάβει το λόγο. Από ό,τι φαίνεται όχι. Α, και όμως, ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ένα σύντομο σχόλιο από τη Γενική Διεύθυνση Αστικής Πολιτικής. Εμείς χαιρετίζουμε τα σχόλια που εκφράστηκαν εδώ και ε, φιλοδοξούμε στο έκτο πρόγραμμα συνοχής να εξετάσουμε ορισμένα από αυτά τα θέματα. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να μετρήσουμε ποσοτικά την κρίση. Αυτό είναι δύσκολο. Δεν έχει ξεπεραστεί ούτε η ύφεση ούτε η φτώχεια. Η έκτη έκθεση συνοχής θα καλύψει όλα αυτά τα θέματα και μετά από αυτή την έκθεση αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια είναι να συνεχίσουμε να εξερευνούμε πόσο έχουν υποφέρει οι πόλεις από την κρίση και πόσο θα υποφέρουν και κατά τα επόμενα έτη. Είσαστε συγκινείς μιας κυρίας που είναι αθλήτρια. Καλώς. Τελειώνει η συζήτηση. 24 Οκτωβρίου στις 12 η ώρα. Ε, θα ψηφίσουμε στις 26 Νοεμβρίου στην Επιτροπή μας. Η Επιτροπή Ρέγγι θα τοποθετηθεί τον Ιανουάριο και κατόπιν θα περάσει το θέμα το Φεβρουάριο στην Ολομέλεια. Αυτά για το σημείο 17. Ε, Στο 18 και εδώ έχουμε έκθεση του κυρίου Κόζα που ε, δεν θα έρθει, αλλά η κυρία Μπάουερ τον ε, αντικαθιστά. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση αυτή συντάχθηκε πάνω σε μια έκθεση που δεν ήταν συνηθισμένη γιατί η έκθεση του Λουί Μισελ δεν ακολουθεί την ε, συνηθισμένη διαδικασία. Είναι το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον, δηλαδή πώς θα αλλάξουν οι συνθήκες ε, με τι νέες πτυχές, ε, με τι τρόπους συνεργασίας με το Συμβούλιο. Είναι μέτρα θεσμικού χαρακτήρα. Και στο δεύτερο μέρος της έκθεσης αναφέρονται οι αρχές της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης. Δεν μιλάει για αδελφότητα, μιλάει και για την ηθογένεια και την δικαιοσύνη. Δεν είχαμε ακόμα την ευκαιρία να έχουμε πάρει αυτή την έκθεση γιατί η έκθεση πηγαίνει πέρα από τις δυνατότητες που μας προσφέρει η συνθήκη. Η γνωμοδότηση αυτή έχει να κάνει με τη σημερινή κατάσταση και σύμφωνα με τον κύριο Κόσα το σχέδιο αυτό που θα έπρεπε να συζητηθεί στην Επιτροπή μας χρειάζεται να συμπεριλάβει και κοινωνικά στοιχεία κοινωνικής πολιτικής σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Επιτροπή Απασχόλησης πρέπει να συντάξει μία έκθεση με λεπτομέρειες και συμμερίζομαι την άποψη αυτή Νομίζω ότι η Επιτροπή μας είναι η αρμόδια Επιτροπή πάνω σε αυτό το δύσκολο θέμα γιατί κυριαρχεί ένα δίλημα. Είναι ένα θέμα για το οποίο δεν έχουμε βρει ακόμα λύση αλλά νομίζω ότι οι συνάδελφοι συμμερίζονται αυτή την άποψη. Να ζητήσω κάτι από τους συναδέλφους να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε κοινωνικά θέματα, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εργασία και την απασχόληση, γιατί αυτό είναι το κύριο έργο μας. <laughs> Az a nagy Ναι, αυτά λοιπόν. Έχω την τιμή να ζητήσω από τους συναδέλφους αν έχουν κάποια ερώτηση να υποβάλουν ή κάποιο σχόλιο. Ποιος θα επιθυμούσε να λάβει τον λόγο, ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάξει, έχετε τον λόγο. Όχι, δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της ομάδας εργασίας μας γιατί δεν γνωρίζουμε το κείμενο και η Βίρη Σίπελ, εξοικειώδης ηγήτρια, ε, θα πρέπει ακόμα να συντάξει τροπολογίες αλλά παρακολούθησα προσεκτικά τα όσα είπες και δεν ξέρω ε, σχετικά με αυτό που λέει και ο Κώσα δηλαδή το ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε ιδιαίτερα την προσοχή μας τα κοινωνικά δικαιώματα τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα αυτή θα είναι και η στάση δική μας είναι η προστιθέμενη αξία που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε σε αυτή την έκθεση, να δούμε μέσα από αυτή την προοπτική αυτή την Επιτροπή μας αυτό και θα κάνουμε, δεν έχουμε στη... Δεν έχουμε τις μεταφράσεις, αλλά θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας, επαναλαμβάνω, σε αυτό. Και για να το πει στον Κώσσα, το σημαντικό είναι να δει κανείς κάτι που είναι κανονικά κρυμμένο, κρυφό. Μιλάει για τα θεμελιώδη δικαιώματα για να μιλώντας για τα ατομικά δικαιώματα αλλά είναι εδώ η κοινωνική διάσταση αυτών. Υπάρχουν και τα συλλογικά δικαιώματα που είναι και αυτά θεμελιώδη. Τους συνεταιρίζεστε για την ε, απεργία κλπ. Και αυτό είναι ο συλλογικό χαρακτήρα. Αυτό είναι δεύτερο. Ε, και υπάρχουν και τα αυτόνομα, όπω είπαμε, τα αμεμονωμένα. Και τα ατομικά και η συσολιστική ομάδα θα επωφεληθεί από αυτή την έκθεση Κόσα για να τα πει αυτά τα πράγματα που δεν έχουν αναφερθεί, δεν έχουν τεθεί ανάγλυφα. Υπάρχουν πάρα πολλά εκατομμύρια εργαζόμενοι που δεν μπορούν να προσ... που, που προστατεύονται συλλογικά αλλά και μεμονωμένα όμως εξαρτώνται από και κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και από ακραία φτώχεια. Αυτά είναι ουσιαστικά τα στοιχεία τα οποία η σοσιαλιστική ομάδα θα προσπαθήσει να υποστηρίξει και εποφελούμε από τα τελευταία δευτερόλεπτα που είναι εδώ. Πρόεδρος, για να δούμε αυτό το φιλελευθερισμό. Λοιπόν, θα μας ακούσουν ε, θα μας ακούσει και θα εισακούσει και την άποψη των σοσιαλιστών τη θέση μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την κατανόησή σας. 24 λοιπόν Οκτωβρίου, 12 η ώρα, είναι η προθεσμία και ε, στις 5 ε, Δεκεμβρίου θα ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό και στις 5 ε, Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε. Η κυρία Μπάουερ έχει τον τελευταίο ε, λόγο. Μια πρόταση, αν μου επιτρέπετε, το, σχε... το του σχεδίου της γνωμοδότησης είναι στο EPNet εδώ και αρκετό καιρό και σε διάφορες γλώσσες. Ίσως να μην το βρει και ο σκιώδης σας. Το Τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι το 22. Εδώ λοιπόν μιλάμε για το θέμα διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο ε, FEAD, η κυρία Κοστέλο, ο κύριος Αλεσάνδρο θέλει να πει κάτι πολύ σημαντικό. Αλεσάνδρο, έχεις το λόγο. Ναι, η κυρία Κουστελού έπρεπε να αποχωρήσει γιατί είχε προβλήμα με την πτήση της και μου άφησε ένα μικρό σημείωμα ενημερώνω, ενημερώνοντάς με για το αποτελέσμα των διαπραγματεύσεων χθες το βράδυ και για τις αποφάσεις που έλαβε το Συμβούλιο για αυτό το Ταμείο για τη βοήθεια προς τους άπορους. Βασικά είναι καλά τα νέα γιατί ουσιαστικά συνάδουν με τις ανησυχίες αυτές της Κομισιόν καταρχήν Πρέπει να πούμε ότι οι επιλές που υπήρχαν για το ταμείο αυτό δεν υλοποιούνται, δηλαδή θα συνεχίσει να υπάρχει ένα ταμείο που είναι τόσο σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες, ε, που είναι άποροι, δεν έχουν ούτε καν τρόφιμα και τα άλλα σημαντικά θέματα που σχετίζονταν με τη δική μας Επιτροπή. Για τα θέματα αυτά θα υπάρχει ένα μείγμα μεταξύ της συμμετοχής όλων των κρατών μελών και θα έχουμε και ένα εκούσιο τμήμα. Όμως ε, γενικά τα μεγέθη ικανοποιούν όλες τις απόψεις που εκφράστηκαν σε αυτήν την Επιτροπή. Όλες οι χώρες θα συμμετέχουν στο επίπεδο του 3,5 δισεκατομμυρίων και θα υπάρχει και ακόμα ένα έξτρα δισεκατομμύριο για όσους εκούσια επιθυμούν να το χορηγήσουν. Επίσης ε, κ. Κοστελό θεωρεί ότι προχωρούμε σε ικανοποιητικούς ρυθμούς ε, προκειμένου να αναλάβουν το όλο που τους αξίζει όλοι οι εταίροι για να εξυπηρετήσουν τους στόχους του Ταμείου. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα και ίσως θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση γι' αυτό στις επόμενες συνεδριάσεις. Υπάρχει επιθυμία από το Συμβούλιο να επεκτείνει το ταμείο να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογή του τομείου και να καλύπτονται και άλλες δραστηριότητες. Και εδώ, ξέρετε, έχουμε τον κοδόνα του κινδύνου, γιατί ουσιαστικά έμεσα το Συμβούλιο προσπαθεί να λιώσει ε, την, το τρόπο εφαρμογής αυτού του ταμείου και ότι καλύπτει τους πιο άπορους Και ουσιαστικά εδώ μιλάμε για την παροχή των πιο βασικών ε, υλικών αγαθών ε, για την επιβίωση. Και γι' αυτό ε, υπάρχει επιφύλαξη από την πλευρά της ηγήτριας και θα επανέλθει στα θέματα αυτά και να ενημερώσει την Επιτροπή. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αλισάνδρο είναι αγγελιαφόρος καλών ειδήσεων, πολύ ωραία, και κυρίως ε, η ευρωπαϊκή υπεραξία. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ε, Σάμπα, έχετε το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε ο συνάδελφος και εγώ συμμετείχα χθες στον τριμερή διάλογο να σας πω μερικά πράγματα. Δεν είμαστε εδώ πολλοί παρόντες, αλλά να πούμε στα πρακτικά το εξής. Οι συνθήκες εργασίας είναι απαράδεκτος εδώ. Γιατί ξεκινάμε τις εργασίες μας στις 8 το βράδυ για τον τριμερή διάλογο και δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε για μακρύ χρονικό διάστημα, γιατί είμαστε πολιτικοί, εντάξει, είμαστε συνηθισμένοι σε παρόμοια εργασίες, αλλά έστω και να αντιδράμε δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό και είχαμε και τους διερμηνείς που ήταν γιατί αν ήταν ας πούμε διερμηνείς από τις 8 το πρωί μέχρι τότε το βράδυ δεν θα μπορούσαν εκείνοι να δουλέψουν. Και χθε το βράδυ εντάξει δεν είχαμε, δεν διαθέταμε διερμηνία μας είπαν ότι δεν υπήρχαν αρκετοί διερμηνείς για να μας καλύψουν αλλά εγώ δεν ξέρω αγγλικά και για μένα χωρίς διερμηνία ήταν δύσκολο. Δεν είπα ότι δεν κατάλαβα και τίποτα από όσα είπαν οι συνάδελφοι, το κάτι της μου το κατάλαβα. Εδώ συμφωνώ με όσα είπε λοιπόν ο προηγούμενος ομιλήτης τι με ανησύχησε κάπως ε, οι προϋποθέσεις για την ε, ε, συμφωνία στο Συμβούλιο θα πρέπει να τις δούμε. Εδώ δεν θα ήταν μόνο για τους περισσότερο άπορους όσον αφορά τροφή, αλλά επίσης και μια συνθήκη κοινωνική η οποία αντιμετωπίζεται υπό την ευρύτερη της έννοια και με μια θα δούμε και την υποχρεωτική συμμετοχή τι κάνουν προσπαθούν όλοι να συμμετάσχουν εκεί στο ταμείο αυτό αλλά θέλουν να προχωρήσουν και σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτού του ταμείου. Είναι πράγματα δύσκολα. Πρέπει να πετύχουμε μία λύση. Επιθυμούμε να είναι εργαλείο το ταμείο αυτό για, τους, ε, για όσους έχουν περισσότερη ανάγκη. Εντάξει, και από τις 31 Δεκεμβρίου μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να καταργηθεί κιόλα. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά στον επόμενο τριμερή διάλογο. Πράγματι, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ε, νομίζω ότι σχεδόν τελειώσαμε. Θέλω να σε επισημάνω ότι στα διάφορα δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις και η επόμενη συνάντησή μας είναι στις 5 Νοεμβρίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που τελειώσαμε τελικά και πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο. Αυτό δείχνει ότι είσαστε πειθαρχημένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους διερμηνείς. Γεια σας.